So, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίσατε στην ε, συνεδρίαση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής που οργανώνει η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Να καλωσορίσω τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Να σας υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή μας, η ΕΚΟΝ, ήταν ιδιαίτερα δραστήρια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι μεταρρυθμίσεις της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνοδεύονται από αυξημένη δημοκρατική λογοδεσία. Δηλαδή, θα υπάρχει λογοδεσία και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι ιδιαίτερη χαρά να σας υποδεχόμαστε εδώ σήμερα και να ακούσουμε τη συνεισφορά σας σε αυτή τη διακοινοβουλευτική ε, συνεργασία για να ενισχύσουμε το ρόλο των κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οικονομική διακυβέρνηση. Όπως γνωρίζετε, η συνεδρίαση αυτή ε, χωρίζεται σε δύο συνεδρίες. Η πρώτη είναι μια ε, παρακολούθηση των συστάσεων χώρα και το δεύτερο είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εδώ και τον εκπρόσωπο του Ολλανδικ... της Ολλανδικής Γερουσίας που θα συμπροεδρέσει εδώ μαζί μου και είναι και ο κύριος Μάρτιν Φανροχέν... από την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων του Ολλανδικού ε, της Ολλανδικής Γερουσίας που θα συμπροεδρεύσει στο δεύτερο τμήμα της συνεδριασής μας. Επίσης να σας ενημερώσω ότι επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός ε, συμμετοχών κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι ε, δυνατό να λάβετε όλο το λόγο, θα δοθεί προτελειότητα να δώσουμε το λόγο σε όσο το δυνατόν περισσότερες βουλές. Όποιος λαμβάνει το λόγο θα παίρνει το λόγο για δύο λεπτά το πολύ. Ε, θα έχουμε περίπου 20 με 25 παρεμβάσεις δηλαδή και φυσικά θα προσαρμόσουμε και το πρόγραμμα ανάλογα με την εξέλιξη της συζήτησης. Επίσης να σας πω ότι υπάρχουν κάρτες για να ζητήσετε το λόγο. Μπορείτε να συμπληρώσετε λοιπόν το έντυπο. θα ε, τα συμπληρώσετε. Θα προσπαθήσουμε φυσικά να ε, δώσουμε το λόγο αντίστοιχα και σε ευρωβουλευτές και σε βουλευτές, αλλά φυσικά θα προσαρμοστούμε και ανάλογα με την εξέλιξη της συζήτησης. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη τη συνεδρία, παρακολούθηση για τα BEPS, διάβρωση της βάσης και ε, μετατόπιση του χρέους να σας πω ότι είναι η τρίτη φορά που γίνεται κοινή συζήτηση στον τομέα της φορολόγησης. Ε, πριν από δύο χρόνια συζητήσαμε το σύστημα ΦΠΑ και πέρσι συζητήσαμε μια κοινή προσέγγιση για την τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, κυρίως μετά από την αποκάλυψη των του σχεδιασμού για την επιθετική φορολόγηση, τα λεγόμενα Leaks. Έχουν εξελιχθεί πολύ τα πράγματα την τελευταία μας συζήτηση. Ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες ε, ε, με τις συστάσεις για την καταπολέμηση των ΠΕΠΣ e και πριν από δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγής και παρουσίασε και το σχέδιο για τις εκθέσεις αναχώρα για ε, τις ε, πολυεθνικές δράσεις μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών. Θα γίνει λοιπόν αυτή η συζήτηση τώρα και θα μιλήσουμε ως ε, νομοθέτες στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και θα δούμε τις βασικές συστάσεις και την οδηγία BEPS και το πώς μπορεί να μεταφερθεί αυτή στο εθνικό δίκαιο και να καλωσορίσω και τον Αλένα Μασούρ, ο οποίος είναι ε, πρόεδρος της ειδική Επιτροπής ε, Τάξε, η οποία εργάζεται επισταμένα και δίνει ιδιαίτερη όθεση στις δραστηριότητές μας στον τομέα αυτό. Επομένως, όπως ε, θα γνωρίζετε, έχουμε μία ad hoc επιτροπή, η οποία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο θέμα αυτό και θα εξετάσει ε, φυσικά θέματα τα οποία έχουν σχέση και με την ομοθεσία της ε, Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ. είναι χαρά επίσης να έχουμε εδώ και την κυρία, τον κύριο Βαλέρ Μουταρλιέ, ο οποίος είναι διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Ταξιούτζ, την κυρία Κάρολιν Μάλκομ, η οποία είναι από το Κέντρο Φορολογικής Πολιτικής και Διοίκησης του ΟΣΑ. Να ξεκινήσουμε, θα δώσω το λόγο δεν ξέρω αν ο συνάδελφος θέλει να πει δύο λόγια πριν ε, ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο στους περισσότερους από εσά, αλλά φυσικά αυτό θα γίνει αφού ακούσουμε τους ομιλητές ε, και κάνουν τις εισαγωγικές τους παρεμβάσεις. Και εγώ προσβλέπω στη συζήτηση και εκ μέρου ε, τη κοινοβουλευτική ε, διάσταση τη Ολλανδική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και συνδιοργανώνω αυτή τη συνεδρίαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά να σα δώσω το λόγο τώρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρώτο ομιλητή λοιπόν είναι η Καρολίν Μάλκομ από το Κέντρο Φορολογική Πολιτική και Διοίκησης του ΟΣΑ. Δέκα λεπτά έχετε στη διάθεσή σα, Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που με απευθύνατε. Είναι πολύ επίκαιρη στιγμή όπως είπατε για να συζητήσουμε την εφαρμογή των BEPS. Τον Οκτώβριο είχαμε το πακέτο των G20 και του ΩΣΑ για τα πακέτα BEPS για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών και τώρα περνάμε στην εφαρμογή. Πριν όμως αναφερθώ στο ίδιο το πακέτο θα άξιζε ίσως να δούμε γιατί ήταν τόσο κρίσιμο το BEPS για να προχωρήσουμε όσον αφορά τις διεθνείς ε, φορολογικές ε, διευθετήσεις και τους φορολογικούς κανόνες και να προχωρήσουμε στον 21ο αιώνα. Μία βασική αρχή μας λοιπόν ήταν πώς θα διασφαλίσουμε σε μία σύγχρονη οικονομία του 21ου αιώνα ε, η δημιουργία του, της αξίας ε, θα ευθυγραμμίζεται με την φορολογία. Γιατί λοιπόν ήταν το σημαντικό αυτό. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν να έρθουν και τα, 20, τα μέλη των G20 και του ΩΣΑ σε μια συνεδρίαση ισότιμη για να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα. Αποφασίσαμε λοιπόν πέρα από το πλαίσιο του ΩΣΑ να δούμε το παγκόσμιο πλαίσιο γιατί αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν μια αναντιστοιχία μεταξύ των ρόλων διαφόρων χωρών και επίσης ε, να ενημερώσουμε και τους διεθνείς κανόνες έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν με τη σύγχρονη οικονομία. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο είχε μεγάλη συμμετοχή και ήταν η πρώτη φορά που εργάστηκε κατά αυτόν τον τρόπο ο ΩΣΑ και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να επιτύχουμε συνένεση στις ε, δράσεις, 15 δράσεις, στις 44 χώρες που εμπλέκονται. Ταυτόχρονα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα βεβαίως, γιατί αυτό το οποίο συχνά ακούμε ως κριτική τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι πως ε, είναι περίπλοκο, περίπλοκο είναι δύσκολα τα συστήματα και περίπλοκα ούτως ή άλλως όσο έχουν. Αλλά η εναλλακτική απέναντι στον ΠΕΠΣ e δεν ήταν να διατηρηθεί το status quo. Η εναλλακτική ήταν ότι κάθε χώρα θα ακολουθούσε τον δικό της ε, δρόμο για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ ακαθόδες ε, πολιτικά, ήταν ιδιαίτερα και από το 2012. Οπότε μας δόθηκε η δυνατότητα μέσω του BEPS να δούμε ακριβώς το ζήτημα των παραθυρακίων που επιτρέπουν την ε, φόρο αποφυγή με έναν τρόπο συνολικό και παγκόσμιο. Μία άλλη σημαντική πτυχή ήταν ακριβώς το ότι είχε μια μορφή διαβούλευσης. Οπότε δεν ήταν μόνο οι 44 χώρες οι οποίες ε, ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη των κανόνων, αλλά έγινε και μια διαβούλευση με 120 συγκεκριμένα χώρες ε, σε περιφερειακές ε, διαβουλεύσεις ε, και άλλες 14 χώρες που ενεπλάχισαν άμεσα και αντικατοπτρίζουν όλο το φάσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Ήταν λοιπόν κάτι το σημαντικό, ήταν ευρύτατη η συζήτηση και εκτός όσα. Επίσης είχαμε πολύ έντονες διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών και νομίζω πως ε, οι προσπάθειες αυτές θα αποδώσουν τώρα που περνάμε στη φάση της εφαρμογής γιατί οι επιχειρήσεις είχαν εμπλακεί, διαμόρφωσαν τα μέτρα έτσι ώστε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του βάρους της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας. Και τέλος, πριν στραφώ στο ίδιο το πακέτο, να αναφέρω πόσο ευρύ είναι αυτό το πακέτο. Πολλοί από τους τομείς που μας απασχόλησαν ε, καλύπτουν ζητήματα που είχαν απασχολήσει τον ΩΣΑ, παραδείγματος χάρη το transfer pricing, φορολογικές ε, συνθήκες, επίσης ε, και άλλους τομείς που περιέχονται στο πακέτο φόρο αποφυγής που είδαμε τον προηγούμενο μήνα εγχώρια μέτρα, παραδείγματος χάρη το κατά πόσον αφαιρούνται οι φόροι, οι Τόκι, με συγχωρείτε. Ή τι γίνεται με θηγατρικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, ενώ οι χώρες παραμένουν κυρίαρχες στα φορολογικά ζητήματα, γεγονός είναι πως είναι δύσκολο να υπάρχει ένα αποτελεσματικό εγχώριο φορολογικό σύστημα χωρίς να λαμβάνει υπόψη το τι συμβαίνει διεθνώς. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά από όλα τα μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Επιτροπή Φορολογικών Θεμάτων και τώρα που έχει ολοκληρωθεί το πακέτο έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση όπως είπα στην, της εφαρμογής και εκεί θα ήθελα να εστιάσω σήμερα. Και ένας χρήσιμος τρόπος να το δούμε αυτό το πακέτο και τα 15 μέτρα είναι να το δούμε ανα ομάδες μέτρων και έτσι ίσως θα βοηθηθούν και οι νομοθέτες για να δουν τις προτεραιότητες, την ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να γίνει η εφαρμογή και ελπίζω να σας βοηθήσει αυτό. Λοιπόν, τι περιέχεται σε αυτό το πακέτο. Πρώτα απ' όλα είχαμε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές, τέσσερις που συμφωνήθηκαν και συμφώνησαν οι χώρες ότι εάν δεν υπήρχε κάποια κοινή δράση θα είχαμε αρνητικές επιπτώσεις σε άλλες χώρες. Τι μιλάμε λοιπόν. Εκθέσεις αναχώρα επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές. Μιλάμε δηλαδή για ανταλλαγή φορολογικών συμφωνιών και προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα. Κατάχρηση φορολογικών συνθήκων όπου καταλήξαμε σε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για το να μην μπορεί κανείς να επιλέγει φορολογικές συνθήκες. Και τέλος, ε, επίλυση διαφορών, γιατί παρά το ότι η BEPS επικεντρώθηκε κυρίως στο ότι δεν θα υπάρχει διπλή μη φορολογία, έπρεπε να δούμε και τις περιπτώσεις διπλής φορολογίας ε, οι οποίες ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είχαμε κατόπιν και ενημέρωση των υφιστάμενων προδιαγραφών, ιδιαίτερα οι κατευθυντήριες γραμμές για το transfer pricing, τη μεταφορά κερδών και βεβαίως ε, κάποια άλλα πράγματα όπως η έννοια της μόνιμης έδρας. Και μετά καταλήξαμε σε κάποιες κοινέ προσεγγίσεις που αφορούν τομείς ε, εργασίας ε, στους οποίους οι χώρες δεν είναι υποχρεωμένες να λάβουν μέτρα, αλλά εάν λάβουν μέτρα θα ακολουθήσουν τα συμφωνημένα. Παραδείγματος χάρη ε, αυτό αφορά τον κανόνα για το αν εκπίπτουν οι τόκοι. Και τέλος, καταλήξαμε σε κάποιες βέλτιστες πρακτικές που ήταν νέος τομέας εργασίας για τον ΩΣΑ ειδικά όσον αφορά τους κανόνες και την υποχρεωτική αποκάλυψη φορολογικών συμφωνιών κάτι το οποίο μας έδωσε μια εικόνα του τι κάνουν οι χώρες αυτή τη στιγμή και προετοιμάζει βεβαίως και τη μελλοντική μας εργασία. Προφανώς κάναμε πάρα πολύ δουλειά για την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας που θα συνεχιστεί στο μέλλον και θα συνεχίσουμε και με τα πολυμερή μέσα. Λοιπόν, θα σταματήσω τώρα εδώ για να περάσουμε στην εφαρμογή. Να σας πενθυμίσω λοιπόν τέσσερις τομείς εργασίας, οι ελάχιστες προδιαγραφές, ε, τέσσερις που θα αποτελέσουν ε, το κύριο μέρος της επόμενης φάσης μας, όπου θα δούμε πώς εφαρμόζουν οι χώρες αυτά τα μέτρα και θα τους βοηθήσουμε στην εφαρμογή. Μετά, Έχουμε ενημέρωση των υφιστάμενων προδιαγραφών, κοινή προσέγγιση και βέλτιστες πρακτικές. Προς τα που πάμε λοιπόν από εδώ και μπρος. Σκοπεύουμε να στηρίξουμε τις ε, χώρες στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, να αναπτύξουμε πρακτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και εργαλεία ε, που στοχεύουν σε λιγότερο ανεπτυγμένες ε, χώρες, όπου ίσως πρέπει να προσαρμοστεί η εφαρμογή των κανόνων δεδομένων των περιορισμένων δυνατοτήτων των χωρών αυτών, αλλά και να παρακολουθούμε την εφαρμογή των τεσσάρων αυτών ελάχιστων προδιαγραφών από τα κράτη-μέλη και να συνεχίσουμε βεβαίως με την, το τεχνικό σκελό της εργασίας μας. Λοιπόν, πηγαίνουμε τώρα στο συνολικό πλαίσιο, το οποίο έχει στόχο να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής πέρα από τις 44 χώρες που έχουν εμπλακεί μέχρι στιγμή για να έρθουν και άλλες χώρε στο πακέτο αυτό. Ήταν μια αρχή μας ότι θα πρέπει να είναι παγκόσμιοι αυτοί οι κανόνες και θα προσκαλέσουμε χώρες στην επόμενη φάση να συμμετάσχουν ισότιμα με τα μέλη του ΩΣΑ και του G20 που είναι ήδη μέλη και βέως ο ρόλος θα είναι να υπάρξει μια παρακολούθηση της ε, εφαρμογής, να αναπτύξουμε την ε, στήριξη των δυνατοτήτων των χωρών για την εφαρμογή και βεβαίω να δοθεί συνέχεια στο τεχνικό σκέλος. Όσον αφορά λοιπόν τώρα την εφαρμογή, αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα εργαστούμε ως με τους G20 και ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε επόμενες φάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στην Βαλερή Μουτουαλιέ από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακαλώ στον κύριο Βαλερή ο κύριος Βαλερή Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε και κύριοι βουλευτές χαίρομαι που για δεύτερη φορά συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση όσον αφορά την φορολογική βελτιστοποίηση είμαι διευθυντή, λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τμήμα που ασχολείται με τη φορολογία. Θα προσπαθήσω μην επαναλάβω αυτά που μόλις ανέφερε η Καρολίν γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος. Κίνδυνος να επαναληφθούμε επειδή το θεματολόγιο μας σε επίπεδο ένωσης είναι θεματολόγιο εφαρμογής. Δηλαδή εξετάζουμε τα αποτελεσμάτα των συζητήσεων που γίνονται γενικά και προσπαθούμε να συντονίσουμε την εφαρμογή τους στην εσωτερική αγορά ώστε αυτό να γίνεται με τρόπο συνοπή και να, προσθέτουμε, και να προσφέρουμε ένα πλαίσιο κανονιστικό και νομοθετικό θετικό για τις επιχειρήσεις. Να μιλήσω λοιπόν για το περιεχόμενο των προτάσεων και για την μέθοδο που ακολουθούμε για να προχωρήσουμε στην εσωτερική αγορά και τις εταιρικές σχέσεις που χρειαζόμαστε βέβαια αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας δηλαδή να αποτελέσουμε ένα πιο σωστό πλαίσιο όσον αφορά την κατανομή του φορολογικού φόρτου στην εσωτερική αγορά, αλλά που ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι και ελκυστικό για τι επιχειρήσει. Όσον αφορά λοιπόν το πεδίο που καλύπτουν οι δράσει μα, νομίζω ότι δεν ε, σφάλω λέγοντα ότι το σύνολο των στόχων και των δράσεων που έχουν εντοπιστεί συνολικά από το BEPS αντανακλώνται και μεταλαβαδίζονται στην Ένωση. Νομίζω ότι για μας αυτό είναι ένα θέμα αξιοπιστίας. Δηλαδή θέλουμε να αποτελέσουμε σε επίπεδο G20 ένα εταίρο ο οποίος είναι ένεργος σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το θεματολόγιο και είναι και ένα θέμα, και ένα θέμα αποτελεσματικότητας γιατί προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε αυτές τις προδιαγραφές με τρόπο συντονισμένο στην ενιαία αγορά, ώστε να έχουμε περισσότερη ευκολία για τις ε, χώρες μας όσον αφορά την ε, δημιουργία της φορολογικής βάσης αλλά και για την ασφάλεια δικαίου για τους φορολογικούς οικονομικούς φορείς. Είναι και ένα θέμα φορολογικής ισότητας επίσης και δικαιοσύνης γιατί είναι αλήθεια ότι η αρχή φορολόγησης ε, στην πηγή των κερδών ε, θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην είναι ευλαβερός και για την ανταγωνιστικότητα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά λοιπόν στο θεματολογιό μας. Κάποια γρήγορα παραδείγματα σε σχέση με αυτά πάνω στα οποία εργαζόμαστε. Παραδείγματο χάρη, αυτό που λέμε το pay box, δηλαδή το σχήμα που αφορά την καινοτομία και την έρευνα, που ήταν αντικείμενο δέσμευση όσον αφορά το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών πέρσι όσον αφορά δηλαδή την προσέγγιση σε σχέση με τον ΩΣΑ. Επίσης έχουμε το θέμα της διαφάνειας μεταξύ δημοσίων διοικήσεων, δημοσίων αρχών με την υιοθέτηση της οδηγίας για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων πέρσι ή ακόμα και το πρόγραμμα εργασίας που έχουμε εφαρμόσει όσον αφορά τις μεταφορές, όσον αφορά τα κοινά φόρου μεταξύ διοικήσεων και επιχειρήσεων για την ενημέρωση των τιμών. Και τον Γενάρη προτείναμε και την ε, υποβολή εκθέσεων αναχώρα και αναφορολογική αρχή πάντοτε στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ ήδη έχουμε έτσι μια κυκλομορφία εργαλείων, εργαλείων συγγνώμη, όσον αφορά τα προβλεπόμενα από τον ΩΣΑ για να καταπολεμήσουμε βεβαίως την ε, διαφυγή κερδών μέσω κανόνων που αφορούν τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό, τα ευρωπαϊκά προϊόντα, ε, θέματα όλα αυτά που είχαμε προτείνει στα πλαίσια της οδηγίας για την φορολογική βελτιστοποίηση πριν από δύο εβδομάδες και που θα συμπληρωθούν και από άλλες πρωτοβουλίες όπως ε, για παράδειγμα αυτές που προθέμεθα να κάνουμε σε άμεσο χρονικό διάστημα. Όπως έλεγα προηγουμένως, όλα αυτά συνεχίζονται, μεταδίδονται στις δράσεις μας, συνεχίζοντας βέβαια και με τις εργασίες στα πλαίσια του ΩΣΑ. Τώρα για τη μέθοδο. Έχω μία εργαλειοθήκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας επιτρέπει να εντοπίσουμε το βέλτιστο εργαλείο για να καταλήξουμε στους στόχους που επιθυμούμε. Να διευκρινίσω εξ αρχής το σημείο αυτό και να πω ότι αυτό αφορά τα διασυνοριακά θέματα. Δηλαδή, ο λόγος δράσης μας σχετίζεται βεβαίω με, με το σύνολο της ενιαίας αγοράς και αποβλέπει κυρίως στην αντιμετώπιση θεμάτων στρέβλωσης στην ενιαία αγορά δηλαδή διασυνοριακά ζητήματα. Όσον αφορά την μέθοδο την οποία ακολουθούμε. Αυτή αποβλέπει στην διαφύλαξη τριών αρχών. Καταρχάς η αρχή της κυριαρχίας των χωρών μελών μας όσον αφορά τη χάραξη των αφορολογικών πολιτικών άμεση φορολογήσεις. Δεύτερον, είναι το ζήτημα της ε, τήρησης και σεβασμού αρχής και επικουρικότητας που ε, λέει ότι πρέπει να παρανεύουμε στο καταλληλότερο επίπεδο και μετά η αναλογικότητα, η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τα εργαλεία τα οποία προτείνουμε και τα οποία θέτουμε επιτάπητος προς στο Συμβούλιο μεταξύ των χωρών μελών. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτές τις αρχές και αυτά τα εργαλεία τα οποία προτείνουμε για την υλοποίηση αυτού του θεματολογίου. Βεβαίως έχουμε ένα εργαλείο στη διάθεσή μας το οποίο είναι ένα νομοθετικό εργαλείο. Από τη στιγμή λοιπόν όπου εντοπίζεται ένα κίνδυνος που αφορά τη λειτουργία ή τις ελευθερίες της ε, νέας αγοράς, κάθε φορά πρέπει να ρυθμίσουμε την εσωτερική φορολογική ανταγωνιστικότητα. Τότε προστρέχουμε σε κάποια εργαλεία όπως οδηγίες. Αυτό ακριβώς κάναμε στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας είτε αφορά αυτό ας πούμε αυτόματη ανταλλαγή τραπεζικών δεδομένων είτε αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών δεδομένων όπως ακριβώς προτείναμε πριν από δύο εβδομάδες δηλαδή την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Εδώ πράγματι αποβλέπουμε στο να διασφαλίσουμε ότι οι διατάξεις που θα πρέπει κάθε χώρα μέλος να υιοθετήσει στα πλαίσια της εθνικής της νομοθεσίας θα πρέπει να λαμβάνονται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κατακαιρματισμός της ενιαίας αγοράς και να διαφυλάσσεται η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και η ελευθερία μετεγκατάστασης. Ένα άλλο θέμα αφορά το εξή. Σε τομεί όπου δεν έχουμε προσαρμογή τη νομοθεσία, αλλά κάνουμε σύσταση στις χώρε μέλη για αναθεώρηση των διμερών φορολογικών συμφωνιών, ή με τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποίησε η με τριτε χωρες αυτο ειναι ενα εργαλειο το οποιο χρησιμοποιησε η κομισιον για να κάνει τη σύσταση σε χώρες μέλη για να αναθεωρήσουν ας πούμε την έννοια τη μόνιμη έδρα, ώστε να δυσφαλίσουμε το ότι όταν μια οικονομική δραστηριότητα λάμβανε χώρα σε μια χώρα μέλος θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάλληλη φορολόγηση των κερδών. Τέλος, το τρίτο εργαλείο το οποίο διαθέτουμε και το οποίο χρησιμοποιούμε σε επίπεδο νοσιακό είναι ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών. Γνωρίζετε ότι έχουμε μια ομάδα που αφορά τον κώδικα διατολογία για την φορολόγηση των επιχειρήσεων που αφορά τις χώρε μέλη, οι οποίες διοργάνουν ένα είδο ε, αξιολόγηση ομοτήμων όσον αφορά τα φορολογικά στοιχεία, ώστε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη διαφάνεια, συνέπεια και έλλειψη στοιχείων βλαβερού ανταγωνισμού. Όσον αφορά τώρα τη μεθοδολογία, ξέρουμε ακριβώς τι θα πρέπει να κάνουμε. Έχουμε κάποια εργαλεία τα οποία μας επιτρέπουν να το κάνουμε αυτό και να προοδεύσουμε, να προχωρήσουμε. Για να το κάνουμε αυτό λοιπόν έχουμε εταιρικέ σχέσεις οι οποίες όμως πρέπει να είναι οι σωστές. Ήδη έχουμε μία πρώτη η οποία ήδη έχει εδρεωθεί σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Έχουμε εδώ ένα φυσικό σύμμαχο ο οποίος είναι το Κοινοβούλιο Γι' αυτό ακριβώς το θεματολόγιο δηλαδή της φορολόγησης των επιχειρήσεων. Έχουμε πολύ θετικές συμβολές μέσα από τις ε, εκθέσεις της Επιτροπής ΕΚΟΝ και της Επιτροπής ε, ΤΑΞ που καθορίζουν ένα θεματολόγιο αρκετά φιλόδοξο θα έλεγα επί το οποίο η Κομισιόν βεβαίως θα ασχοληθεί τους ερχόμενους μήνες. Έχουμε επίσης και ένα Συμβούλιο Υπουργών το οποίο βεβαίως η Ολλανδική Προεδρία εξέτασε μάλλον έθεσε το θέμα της φορολόγησης των επιχειρήσεων μέσα στις ε, πιο υψηλέ προτεραιότητες και ε, θα προσπαθήσουμε να το προχωρήσουμε αυτό. Επίσης έχουμε και μια σημαντική εταιρική σχέση με τις χώρες μέλη γιατί τα φαινόμενα που παρατηρούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε να υπάρχουν και σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι επειδή ακριβώ έχουμε αύξηση τη φορολογική πίεση σε σταθερή φορολογική βάση, όπω η φορολόγηση τη εργασία, τώρα όλα αυτά φτάνουν στα όρια του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι πολίτε ότι το σύνολο των φορολογουμένων θα συμβάλλουν το κομμάτι που τους αναλογεί όσον αφορά την φορολογία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε αυτό το θεματολόγιο σε επίπεδο Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη δική σας συμβολή είτε μέσω πίεσης, άσκηση πίεσης στις χώρες σας στα πλαίσια του Συμβουλίου είτε μέσω διασφάλισης της ε, μεταφοράς και ενσωμάτωσης των μαθητικών πράσεων που έχουν εκδοθεί και που έχουν εγκριθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Είναι φιλόδοξο αυτό το θεματολόγιο, γι' αυτό ακριβώς η συμβολή σας είναι πολύτιμη και απαραίτητη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για τον 1,5 λεπτό χρόνο μου παραπάνω που χρησιμοποίησα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στους άλλους δύο ομιλητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα να δώσω το λόγο στον Αλέλα Μασούρ, τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Τάξε. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε το θέμα αυτό της φορολόγησης των επιχειρήσεων μέχρι πριν από 1,5 χρόνο θεωρούνταν ένα τεχνικό και ανιαρό ζήτημα. Μετά είχαμε τα LuxLeaks, τα οποία ήρθαν να προσθεθούν σε αντίστοιχες αποκαλύψεις του είδους και ξαφνικά σε κάθε χώρα μας έγινε ένα πολιτικό πρόβλημα ε, πρώτης γραμμής ε, και στην Ευρώπη αλλά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ε, έχουμε εδώ και βουλευτές από το Κεμπέκ και είμαστε σε επαφή και με το Κογκρέσο στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό το οποίο ε, προκύπτει είναι ότι τα LuxLeaks θα σημειώσουν μια, ένα τέλος εποχής και μια αλλαγή εποχής ε, στην υπόθεση των LuxLeaks, ε, της φορολογίας των επιχειρήσεων. Θα υπάρχει ένα πριν και ένα μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει άμεση αρμοδιότητα σε θέματα φορολόγησης. Ε, εσείς, ε, οι εθνικοί βουλευτές, ε, είναι, είστε αυτοί που έχετε τον πρώτο αλλά και τον τελευταίο λόγο. Έχουμε παρόλα αυτά καθήκον καταρχάς να ασχοληθούμε σε επίπεδο πανευρωπαϊκό για να δούμε τι πρακτικές υπήρχαν και δεύτερον πρέπει να κάνουμε συστάσεις οι οποίες θα συμπληρώσουν και θα επιβεβαιώσουν ε, τις πρωτοβουλίες οι οποίες ελήφθησαν ε, σε επίπεδο ΩΣΑ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι έρευνές μας ε, κατέδειξαν τρία πράγματα. Πρώτον, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα φορολογικά μας συστήματα στις επιχειρήσεις δεν είναι προσαρμοσμένα ε, στον 21ο αιώνα. Ξεκίνησαν πριν από 100 χρόνια και δεν έχουν προσαρμοστεί στην παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων, στην παγκοσμιοποίηση της διαδικασίας παραγωγής, στην ε, παγκοσμιοποίηση του τρόπου χρηματοδότησης και επίσης ε, στις καινοτομίες που έχουν προκύπτει από την ψηφιακή οικονομία και τον ψηφιακό κόσμο. Δεύτερη διαπίστωση, οι επιχειρήσεις αυτές, οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις ε, καταφέρνουν να ε, αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και στα επίπεδα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια μεγάλη πολυεθνική σε μια απομονωμένη ίσως και μικρή χώρα. Τρίτη διαπίστωση, ακόμα και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μέχρι πρόσφατα ε, χάναμε ε, φορολογικά έσοδα από τη μία χώρα στην άλλη. Ο καθένας από εμά είναι ο φορολογικός παράδεισος κάποιου άλλου. Και εμείς ε, κάναμε συστάσεις στην έκθεση της Λίζα Φερέιρα και του κ. Τόιρερ και προτείνουμε μια συνεκτική φιλισική, να εφαρμόζουμε την επιβολή της φορολογίας, τους κανόνες και τις αρχές του ανταγωνισμού που στην Ευρώπη εφαρμόζουμε σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητε, Δηλαδή τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και την ισοτιμία. Ενώ ε, μέχρι τώρα σε θέματα φορολόγησης επιχειρήσεων ε, υπήρχε ανταγωνισμός ε, ε, χωρίς καμία διαφάνεια, με απόλυτη έλλειψη δικαιοσύνης και χωρίς καμία αξιοπιστία. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία για μας μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουμε την ευρωπαϊκή οικογένεια και θέλουμε να καταλήξουμε στον ίδιο ορισμό για τα φορολογητέα αγαθά σε κάθε χώρα και από αυτή τη βάση θα μπορούσαμε να έχουμε διάφανο και ε, θεμητό ανταγωνισμό στην φορολόγηση. Δηλαδή να φορολογούνται τα αγαθά αυτά ε, όπως γίνεται η φορολόγηση για το ΦΠΑ εδώ και 20 χρόνια και κάτι το οποίο λειτουργεί και σχετικά ικανοποιητικά. Ε, Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουμε και τις συστάσεις του ΩΣΑ, αλλά εδώ θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι μεγάλοι παγκόσμιοι εταίροι μας, ξεκινώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους υπόλοιπους μεγάλους εταίρους, θα συμμετέχουν και αυτοί σε αυτές τις εργασίες και θα συμμερίζονται αυτή τη φιλοσοφία. Το καλό νέο είναι ότι οι πολυεθνικές αρχίζουν να αλλάζουν λίγο στάση λόγω πίεσης από την κοινή γνώμη που εμείς οι εκπρόσωποι, οι αιρετοί του λαού έχουμε ξεκινήσει και οι μεγάλες πολυεθνικές αντιλαμβάνονται ότι όπως δεν μπορούν πλέον να έχουν την πολυτέλεια, να ρηπαίνουν ε, και να κάνουν δραστηριότητες οι οποίες ε, επιβαρύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη, δεν μπορούν επίσης να έχουν την πολυτέλεια να φαίνονται ενώπιον των ε, καταναλωτών τους ως πολίτες που δεν πληρώνουν φορολογία εκεί που δραστηριοποιούνται. Και επίση πρέπει να σα πω ότι η πρόθεσή μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινήσει, να συνεχιστεί αυτή η έρευνα, να εμβαθύνουμε κι άλλου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μετά από τη σημερινή συνεδρία έχουμε προτείνει άλλε δύο διακοινοβουλευτικέ συνεδριάτε, μία στι 16 Απριλίου με του ίδιου συμμετέχοντε και η άλλη στι 2 Μαου στα πλαίσια του ΟΣΑ, καλώντα ε, και τα κοινοβούλια όλων των χωρών που έχει ε, ε, όσα και να πω επίσης ότι ε, προσβλέπω στην αγαστή μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο τώρα το λόγο στον κύριο Μπαγιέ, ο οποίο είναι ο εισηγητή για τα θέματα των ΠΕΠΣ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω και ο συνάδελφο Λαμασούρ, χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να συζητήσουμε και λίγο και τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προέκυψαν μετά από την πίεση ε, της κοινή γνώμης. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι ε, δεν μπορούμε να έχουμε μέτρα χωρίς εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολόγησης. Μία δίκαιη φορολόγηση θα γίνει ο ακρογωνιαίος λήθος της νέας αγοράς. Υπάρχει η μελέτη του ΩΣΑ και η βελτιστοποίηση που γίνεται από τις πολυεθνικές, η επιθετική μάλιστα βελτιστοποίηση οδηγεί σε 4 με 6% απώλειες παγκοσμίως σε φορολόγηση, 40 με 60 δις περίπου δηλαδή ετησίου, πρόκειται για ε, ένα, μια τεράστια απώλεια και αυτό φυσικά θα μπορούσε να βελτιωθεί τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο προτείνει ο Πιέρ Μοσκοβισή στο νέο πακέτο είναι να έχουμε ένα στάδιο το οποίο δείχνει ότι πρέπει ε, να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα των, ε, της των επιχειρήσεων. Όπως είπε και ο κύριο Λαμασούρο, εμεί δεν μείναμε αδρανής, αλλά ε, προχωρήσαμε καταρχάς χάρη στις συστάσεις της έκθεσης του Ρερ Φερέρα και χαίρομαι που έχω εδώ την Ελίζα Φερέρα που είναι συντονίστρια της έκθεσης ε, για το ε, τάξ, συντάκτρια μάλλον της έκθεσης και έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία για τους φορολογικούς παραδόησους και τα φορολογικά ωφέλη μεταξύ κρατών μελών. Νομίζω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταφέραμε να έχουμε κάποια σημαντικά στοιχεία. Καταρχάς σε εθνικό και ε, διεθνέ επίπεδο θα μπορούμε να αναλύουμε τις πολυεθνικέ. Δυστυχώ δεν μας ακολούθησε το Συμβούλιο και έχει βάλει ένα χρονικό όριο 10 ετών Ελπίζω να μπορέσουν αρκετοί βουλευτές να πείσουν τους ε, κυβερνήσεις τους να το ξανασκεφτούν αυτό το ζήτημα, διότι άπαξ και υπάρχει ένα tax ruling θα πρέπει να αναλύεται και να διαβιβάζεται και στα άλλα κράτη-μέλη και δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά γιατί θέλουν να επανέλθουν στο Συμβούλιο με αυτό το όριο των 10 να προβλεφθούν και κυρώσεις. Γνωρίζουμε ότι όλοι θέλουν να είναι καλοί και ευγενεί, αλλά όταν υπάρχουν οι κυρώσεις θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι εφαρμόζονται. Τρίτον, θα θέλαμε το Συμβούλιο Υπουργών να εξετάσει λίγο τα θέματα καλύτερα. Γι' αυτό και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αυξήσει τα καθήκοντά της ως θεματοφύλακας. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, να δημοσιεύονται σαφέστατα όλες τις φορολογικές συμφωνίες των πολυεθνικών. Επίσης να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός αριθμός αναγνώρισης για όλες τις ε, πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και αυτό θα διευκολύνει τα πράγματα και για τις πολυεθνικές αλλά και για τις ε, διοικήσεις. Και επίση υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρότεινε ο ΣΑΚ. Σίγουρα πρέπει να ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, να την ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν και δύο μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, τα οποία θα εξετάσουμε τον επόμενο μήνα. Το θέμα τη ανταλλαγή πληροφοριών ε, για το τι εκθέσει χώρα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα τη φορολόγηση. Και ένα δεύτερο μέτρο είναι οι προτάσει για τα BEPS φυσικά, τα οποία θα σταθώ λίγο, γιατί όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, είμαι ο εισηγητής για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν ε, συγκεκριμένα μέτρα εδώ, η ε, διεύρυνση του, ε, του ελέγχου των ε, πολυεθνικών θα πρέπει η θηγατρική να καταβάλει τους φόρους τους και να μην τους καταβάλει η ε, μητρική εταιρεία που βρίσκεται σε κάποιο φορολογικό παράδοσο και επίσης πρέπει να φροντίσουμε να ε, γίνεται αυτόματη φορολόγηση στη χώρα καταγωγής και να μην υπάρχει φορολογικός παράδεισος ε, στην έδρα που μπορεί να έχει και 40% λιγότερη φορολόγηση. Ξέρετε επίσης ότι οι πολυεθνικές τους ε, έχουν την πνευματική τους ιδιοκτησία σε δικαιοδοσίες που έχουν μικρή φορολόγηση. Αυτό φυσικά αποτελεί μεγάλη απώλεια στις χώρες τις οποίες ξεκίνησε αυτή η πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης υπάρχει το θέμα των επιτοκίων και των φόρων πολύ σημαντικών ε, ε, εκπτώσεων σε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε και ένα γενικό μέτρο της καταπολέμησης των καταχρήσεων. Ε, εγώ πιστεύω ότι λείπουν κάποια ουσιαστικά στοιχεία ώστε να μην διαφεύγουν οι πολυεθνικές και φυσικά θα πρέπει να ε, υποχρεούνται να καταβάλουν φόρες στις χώρες όπου πραγματικά ασκούν μια οικονομική δραστηριότητα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Επίσης, ε, η Google, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι είναι πρωτοπόρος σε αυτές τις πρακτικές, αλλά δεν είναι η μόνη, υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις που ασκούν αντίστοιχη δραστηριότητα. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε όλα αυτά, διότι ξέρουμε όλοι ότι η πολυεθνική, η οποία δεν καταβάλει φορολογία στη χώρα στην οποία ασκεί η οικονομική δραστηριότητα, δεν αποτελεί και υπόδειγμα επιχείρησης. Ε, είναι χρηματοδότηση φορολογία προς όφελος όλων και για την κοινωνική ασφάλεια και για τα έσοδα του κράτους και ούτω καθεξής. Επίσης πρέπει το 2006 να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τα πράγματα για να μειώσουμε το διοικητικό άφθος, το κόστος συμμόρφωσης, ε, την ε, έλλειψη ασφάλειας δικαίου που μπορεί να πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή οι ε, πολυεθνικές για να μπορούν να ε, φορολογούνται βάσει τεχνικού καθεστώτος και φυσικά θα πρέπει να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις να έχουν μία νέα θηρίδα για να αντιμετωπίζουν τα θέματα που αφορούν τη φορολόγησή τους ε, ακόμα και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω όλες αυτές οι πρωτοβουλίε να μην είναι ισμάτιν και ελπίζω το Συμβούλιο να ακούσει τι προτάσει μα. Και θα ήθελα να ε, απευθύνω και μια έκκληση στους παρόντες βουλευτές, διότι εσείς μπορείτε να ασκήσετε πίεση στις κυβερνήσεις σας για να έχουμε πραγματική φορολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα μας αφορά όλους και πρέπει πλέον να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο πρώτος Εθνικού Κοινοβουλίου, ο Δ. Χάνς Μίχελμπαχ από την Γερμανική Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα την χαρά μου για το ότι κατέφεραν οι Υπουργοί Οικονομικών των G20 να καταλήξουν σε μια συμφωνία για την απόκρυψη και την μεταφορά κέρδων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Βεβαίω το σχέδιο δράσης BEPS είναι σωστό, μπορεί να αποτελέσει ορόσημο στην ε, διεθνή πολιτική και στην φορολογική δικαιοσύνη και μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη. Γι' αυτό είναι σημαντικό το ότι το συζητάμε σήμερα. Θα ήταν η πρώτη φορά που θα έχουμε τόσο μεγάλη συνένεση παγκοσμίω για κάποιες παγκόσμιες προδιαγραφές φορολόγησης, κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ποτέ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στα χαρτιά, πρέπει να εφαρμοστεί. Βεβαίως, ο μόνος δρόμος είναι η ε, διεθνής ε, συνεργασία θα πρέπει η βλαπτική ο βλαπτικός φορολογικός ανταγωνισμός ε, και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός να δυσκολέψουν πάρα πολύ. Μεγάλο πρόβλημα βεβαίω αποτελούν οι χώρες οι οποίες δεν έχουν την θέληση ή τα μέσα να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις στις ε, χώρες τους. Ε, το βασικό πρόβλημα λοιπόν ε, το βλέπουμε και σε πολλές συστάσεις που γίνονται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες εφαρμόζονται μόνο μερικώς και με μεγάλη καθυστέρηση. Θα πρέπει όμως τα επόμενα χρόνια να το κάνουν αυτό όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει και περισσότερες χώρες να συνυπογράψουν αυτή τη συμφωνία για να υπάρχουν όσο, το λιγότερο, όσο δυνατόν λιγότερα παραθυράκια και φορολογικές οάσεις. Μόνο έτσι μπορεί το BEPS να λειτουργήσει εις βάθος χρόνου επιτυχώς. Γιατί μέχρι σήμερα οι τίμοι υπεύθυνοι Ευρωπαίοι πολίτες και επιχειρήσεις πληρώνουν περισσότερους φόρους γιατί ακριβώς κάποιες πολυεθνικές επιχειρήσεις ε, μετατοπίζουν και μεταφέρουν τα κέρδη τους αλλού. Πρέπει λοιπόν να το ε, τονίσουμε αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει πλέον στρέβλωση του ανταγωνισμού. Από τη στρέβλωση του ανταγωνισμού δεν κερδίζει καν καμία χώρα σε βάθος ε, χρόνου, ειδικά αν είναι κράτος μέλος της Ένωσης. Βεβαίως, για να επιτύχει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο είναι αποφασιστικό να ε, εμπλακούν και οι ΙΠΑ. Ταυτόχρονα στην εφαρμογή πρέπει να προσέξουμε μην υπάρχει ειδική μεταχείριση για κάποιες χώρες και επιχειρήσεις, ειδικά για τους ε, πρωτοπόρους ε, του φορολογικού dumping, Google, Amazon και λοιπές πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να εμποδιστούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους. Δεν είναι πτέσματα αυτά τα πράγματα, είναι εγκλήματα κατά της κοινή ευημερίας των πολιτών και των υπολείπων επιχειρήσεων. Θα πρέπει επίσης τα μέτρα να εφαρμοστούν ε, ή δυνατόν ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες, αλλιώς πάλι θα έχουμε αυτό το πρόβλημα μεταξύ των χωρών. Δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινήσουν κάποια κράτη-μέλη να τα εφαρμόζουν και να μην το κάνουν οι ΙΠΑ, παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό είναι σημαντικό για εμάς να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας στα εθνικά κοινοβουλία κατά του φορολογικού dumping αλλά και διεθνώς όσον αφορά την φορολογική νομοθεσία και τις ε, πολυεθνικές εταιρείες. Βλέπουμε λοιπόν πως ε, ακόμα δεν υπάρχει μια τέτοια βούληση. Και εδώ πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Σημαντικό λοιπόν, σημαντική πτυχή είναι η αξία να φορολογείται, η προσθέμενη αξία εκεί όπου δημιουργείται. Έτσι νομίζω θα οδηγηθούμε στο, στο δρόμο. Εμείς ή άλλως ε, είμαστε σε μια ομοσπονδιακή χώρα, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και ούτως ή άλλως ισχύει σε εμάς ένα ανάλογο σύστημα, δηλαδή το αφημί για ολόκληρη τη χώρα. Επίσης θα πρέπει να καθοριστούν σαφή όρια για τα patent boxes και να... Υπάρχει εξαίρεση μόνο των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν αναλάβει από μόνες τους την ερευνητική δραστηριότητα. Δεν είναι δυνατόν να την μεταφέρουν εκτός των χωρών με φοροαποφυγή και με, με ευνοϊκή φορολογία. Επίσης θα πρέπει να ισχύει η αρχή οι ίδιοι κανόνες, οι ίδιες προδιαγραφές για όλες τις χώρες, για όλες τις ε, εταιρείε χωρίς εξαιρέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ξεκάθαροι και σαφείς οι κανόνες, γιατί όσο δυνατόν περισσότερο, γιατί όσο περισσότερο περιθώριο ελιγμών υπάρχει, τόσο μεγαλύτερο ο κίνδυνος τρέβλωσης στον Επίσης, Κατά την άποψή μας υπάρχουν κάποια σημεία κριτικής. Αφενός η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε επιβάρυνση ε, των εξαγωγών, να μην υπάρχει δηλαδή διπλή φορολογία και στη χώρα παραγωγής και στη χώρα εξαγωγής. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα πως ε, υπάρχει μία ρήτρα συνένεσης ε, και κάποιες αποκλήσεις σε κάποιες ε, χώρες με κάποια ευρυδικά κατασκευάσματα που αποκλίνουν από τις συστάσεις ε, του ΩΣΑ. Εμείς λοιπόν δεν κατανοούμε αυτές τις αποκλήσεις. Τώρα αν υπάρχουν αποκλήσεις ε, μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ που δεν είναι κράτη-μέλη της Ένωσης, ε, παραδείγματο χάρη ε, με τις ΗΠΑ, θα πρέπει και εκεί πέρα να προσπαθήσουμε να τις αποφύγουμε. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να τελειώσει ο πρόεδρος. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μάρτιν Φανρή από την Ολλανδική Ρωσία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. να συμπληρώσω και να πω ότι ο σανθός δίπλα μου είναι ο κύριος Μάρτιν. Εγώ είμαι Μάνιξ Φανράι. Ευχαριστώ πολύ πάντως εκ μέρους της Ολλανικής Γερουσίας να πω δύο λόγια σε σχέση με πρόσφατες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταπολέμηση της Το πακέτο δηλαδή καταπολέμηση φοραποφυγή που παρουσιάστηκε πριν από δύο εβδομάδες. Αυτό βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Αποτελεσματική φορολόγηση, διαφάνεια και αντιμετώπιση του κινδύνου της διπλής φορολογικής επιβολής, διπλής φορολόγησης. Αφού δημοσίευσε λοιπόν ο ΣΑΤΟ σχέδιο δράσης ε, ΒΑΠΣ στις 5 του Οκτώβρη πέρσι που υιοθέτησε το G20 στις 16 Νοεμβρίου η Κομισιόν πρόθεσε την ατζέντα το θεματολόγιο αυτό Είχαμε το σχέδιο αυτό που συζητήθηκε στην Ολλανδική Γερουσία πρόσφατα. Υποστηρίχθηκαν λοιπόν και οι στόχοι και οι δράσεις του ΠΕΠΣ και προτιμήθηκε η αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με την πιο ήπια. Υπό την άποψη αυτή, η νομοθετική εξουσία της Ένωσης θα είναι προτιμητέα σε σχέση με την πιο ήπια προσέγγιση του ΩΣΑ. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι είχε εκμεταλλευτεί αυτό, αυτή τη συγκυρία προσπαθώντας ακριβώς να μετατρέψει αυτές τις δράσεις ΠΕΠΣ σε σκληρή νομοθεσία και αυστερές συστάσεις. Ο στόχος λοιπόν για την φορά αποφυγή καθορίζει έξι μέτρα για την αποφυγή της. Τα περισσότερα είναι νομίζω το τμήμα του σχεδίου δράσης BEPS, δηλαδή ο κανόνας και η έλεγχη για τις ε, τα υβριδικά, ε, αντικατάχρηση κλπ. Έχουμε επίσης και το switchover, μεταφορά δηλαδή και ε, η οι κανόνες που αφορούν την υπερβολική φορολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα έπρεπε να νομοθετήσει περισσότερο από αυτά που αποφασιστήκαν στο G20 για το πακέτο ΠΑΠΣ. Τα προτινόμενα μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικά και θα πρέπει να τηρούν βεβαίω τι ελευθερίε και τι αρχέ τη επικουρικότητα. Και τέλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ω η νέα αγορά θα έπρεπε να παραμένει μια ελκυστική οικονομία για τους ξένους επενδυτές και για τους επιχειρηματίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγορά θα πρέπει να είναι ελκυστική και ανταγωνιστική σε σχέση με χώρες όπως είπα και στον τομέα της ε, φορολογίας. Το πλεονέκτημα λοιπόν της χλής νομοθεσίας είναι ότι η νομοθετική διαδικασία θα γίνει με τρόπο δημοκρατικό. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο για όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης. Δηλαδή όλες θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτή, αυτές τις οδηγίες, αυτή την νομοθεσία που θα είναι διεθνής και που θα βοηθήσει την Ένωση διεθνώς. Όπως ξέρετε, οι προτινόμενες αλλαγές στην οδηγία για τη διοικητική συνεργασία ακόμα δεν έχουν συζητηθεί στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Το Ολλανδικό Κοινοβούλιο λοιπόν αναμένει μία αξιολόγηση από την κυβέρνηση της Ολλανδίας σε σχέση με τις πιο πρόσφατες προτάσεις. Αυτή τη στιγμή νομίζω αξίζει το να τονίσουμε ότι η υποβολή εκθέσεων αναχώρα ήδη έχει θεσπιστεί από την 1η Γενάρη στην εθνική νομοθεσία. Έχουμε την ενσωμάτωση 13 συστάσεων στην εθνική μας νομοθεσία, κάτι το οποίο αποτεκνύει ακριβώς την ύπαρξη διαφάνειας. Το ίδιο αφορά και τις συστάσεις για τις ε, κοινές προδιαγραφές όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίως θα γίνουν δεκτές από το Κοινοβούλιο, όπως επίσης και οι προτάσεις για την υιοθέτηση φορολογικών αποφάσεων. Τέλος, οι κάτω χώρες υποστήριξαν αναπτυσσόμενες χώρες ώστε αυτές να αναπτύξουν υποδομή φορολογική και προωθήσαμε τη θέσπιση ενός γενικού κανόνα κατά των καταχρήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οπότε ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής το οποίο εστιάζεται στην βοήθεια των αναπτυσσόμενων χωρών σε φορολογικά θέματα θα λάβει βεβαίως μεγάλη υποστήριξη από τη χώρα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάντισλαβ Καμινίσκι τώρα από την Επιτροπή Προπολογισμού του Σλοβακικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την θέση της Σλοβακίας στο σχέδιο ΒΕΠΣ του ωσά Πρέπει να σας πω ότι εμείς αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην σωστή φορολόγηση στη συνεργασία, στην μεταφορά των πληροφοριών και την ενίσχυση των διοικητικών αρχών ώστε να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή και ο σχεδιασμός φοροαποφυγής από τις επιχειρήσεις. Είχαμε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την τεχνική φορολογική νομοθεσία. Είχαμε επίσης και τις κατάλληλες νομοθετικές πρακτικές ώστε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς τη μεταφορά κερδών και την διάβρωση φορολογική ε, βάσης ώστε η φορολογική αρχή μας να είναι σε θέση βεβαίως να κάνει και τους κατάλληλους ε, ελέγχους που αφορούν βεβαίως τις, ε, και τις δυσυνοριακές συναλλαγές. Έχουμε λοιπόν διοικητική συνεργασία που αφορά τα φορολογικά θέματα με άλλες χώρες και η Σλοβακία πραγματικά διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και Θεωρεί η Σλοβακία ότι η πρωτοβουλία BEPS του ΩΣΑ είναι συνεκτική και σημαντική όσον αφορά την αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων στην Ένωση. Η Σλοβακία είναι υπέρ μιας ταχείας εφαρμογής εκ μέρους της Ένωσης των συστάσεων του ΟΣΑ σχετικά με τον ΠΕΠ στην Ένωση επειδή αυτά θα μας βοηθήσουν στο να αποτρέψουμε την ε, μονομερή εφαρμογή από κάθε χώρα μέλη. Θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν όλες αυτές οι προσπάθειες χωρίς να οδηγηθούμε σε επικαλύψεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα Είχαμε πρόσφατα την οδηγία υποβολής έκθεσης αναχώρα η οποία σύντομα θα υλοποιηθεί και η Σλοβακία χαιρετίζει αυτό το πακέτο για την καταπολέμηση φοροαπεφυγής της Κομισιόν που υποβλήθηκε το Γενάρη του 2016. Επίσης, συμφωνούμε με τις ε, συζητήσεις που γίνονται στην Ένωση για αυτό το θέμα και θεωρούμε πραγματικά ότι οι έννοιες του ΠΕΠΣΑ από τον ΩΣΑ θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και θα πρέπει να βοηθήσουν ακριβώ την λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την τήρηση των συνθήκων. Θεωρούμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι εξωτερικέ διαστάσει των BEPS θα πρέπει να εξεταστούν πιο κοντά, πιο στενά και θα πρέπει να αντιδικοποιηθούν οι διάλογοι με τρίτε χώρε ακριβώ για να κυκλοφορήσει για να ε, η έννοια της ε, χρηστής διακυβέρνησης παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον, Έλσικα, στον κύριο Νέλσικα ο λόγος. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε δηλώσεις από τον ΟΣΑ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους προέδρους ε, της Ειδικής ε, Επιτροπής για την ε, Ειδική Επιτροπή για τη Φορολόγηση και από τον εισηγητή για την οδηγία BEPS και ακούσαμε φυσικά και παρεμβάσεις από τρία εθνικά κοινοβούλια, από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σλοβακία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για σύντομες παρεμβάσεις και ερωτήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι έχετε ένα μέγιστο δύο λεπτών χρόνο αργόγορευση. Σας παρακαλώ λοιπόν να έχετε το νου σας το χρόνο και να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Μουέ από την ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για την σημερινή συνεδρίαση ε, διότι είναι η καταπολέμηση της επιθετικής ε, φορολογικής βελτιστοποίησης, διότι χάρη στις προσπάθειες του ΩΣΑ ε, και του G20 η Ευρώπη ασχολείται με το θέμα αυτό. Στη Γαλλία από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα BEPS, εδώ και 3,5 χρόνια έχουμε συστήσει ένα τμήμα ενημέρωσης για το τα θέματα αυτά για να παρακολουθούμε τον ΠΕΠΣ και για να δούμε και τι γίνεται στην εθνική νομοθεσία και σε αυτή την περίπτωση ε, ακριβώς ε, συναντηθήκαμε και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τότε βέβαια στην αρχή ήταν ένα δύσκολο ζήτημα να θίξει κανείς στην Ευρώπη γιατί η φορολογία είναι εθνική κυριαρχία και δεν είχε ακόμα προχωρήσει το θέμα ώστε να φτάσουμε ευτυχώς σε αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Και πράγματι, όπως ε, υπενθύμησαν και κάποιοι, τα LuxLeaks ε, σίγουρα επιτάχυναν τα πράγματα και αποτελούν ε, μια κοινή ανοσυχία πλέον σήμερα όταν μελετούσαμε το θέμα αυτό στην εποχή εκείνη, ξέραμε ότι στην Ευρώπη συμβαίνει το φαινόμενο αυτό και προσπαθούσαμε να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα σφάλματα της εθνικής νομοθεσίας, ώστε να μην μπορούν νομίμως οι πολυεθνικές να μην καταβάλουν φόρους σε καμία χώρα. Και νομίζω ότι το πρόγραμμα των ΠΕΠ e το οποίο υλοποιείται μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δέχεται τις διάφορες προτάσεις. Υπάρχει μια πρόταση ε, που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα και έχει σχέση με την Ευρώπη. Η εναρμόνιση της φορολογικής δάσης ε, για τα, η φορολόγηση των εισοδημάτων των πολυεθνικών και αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν μεν τα επιτόκια, αλλά θα υπάρχουν κοινοί κανόνες που θα ε, διευκολύνουν ε, την ε, ζωή των πολιτών και θα δυσκολεύσουν τη ζωή των πολυεθνικών. Ευχαριστώ. Επόμενος στον κατάλογο ο κύριος Φανρόμπαϊ από την Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κύριε Πρόεδρε, το Βέλγιο συμφωνεί πλήρως με την πολιτική που επιδιώκεται μέσω των BEPS και με τον κύριο Λαμασούρη έχουμε κάποιες επαφές ε, στην ε, Επιτροπή Τάξε για την φορολογία όπου ακριβώς ε, εξετάσαμε κάποια πρωτομησιακά φορολογικά στότα που υπάρχουν με στόχο να προσελκύσουν πολυεθνικές επιχειρήσεις και βεβαίως και τις φορολογικές συμφωνίες ή αποφάσεις και αυτό είναι ένα στοιχείο στο οποίο πρέπει να, δω, να ρίξουμε φως. Και βέβαια έχουμε το γνωστό πρόβλημα του transfer pricing της μεταφοράς των κέρδων. Γνωρίζουμε πως ε, από ευρωπαϊκή πλευρά έχουμε την οδηγία για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων, αλλά Παραδείγματο χάρη ναι, η κυρία Φασταχέρ ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, καταδίκασε το Βέλγιο για το σύστημα αυτό των excessive profit rulings όπως λέγεται μια διπλή μη φορολογία ουσιαστικά και το σύστημα αυτό όμως υπάρχει από το 2004 και με θέλει τώρα να υπάρξει κάποια διόρθωση με τρόπο αναδρομικό και να ζητήσει τα λεφτά πίσω το βελγικό κράτος από τις επιχειρήσεις. Η αναδρομικότητα αυτή ε, της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, δεν ξέρω τι νόημα έχει. Δηλαδή τι νομική βεβαιότητα θα έχει μια επιχείρηση όταν κάνει μια επένδυση και μετά οι ευρωπαϊκές οδηγίες εφαρμόζονται και στην ενδιάμεση περίοδο δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ασφάλεια δικαίου για κάποια φορολογικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο αναφέρθηκε παραδείγματο χάρη για το αν εκπίπτουν οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων, κάτι το οποίο αποτελεί αντικείμενο του BEPS. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σύστημα ονομαστικού τόκου. Άλλες φορές εκπίπτει, άλλες φορές ε, όχι. Τι θα γίνει στην μεταβατική περίοδο τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις διεθνείς εξελίξεις των BEPS ε, και των ευρωπαϊκών οδηγιών. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε να υπάρχει μια νομική βεβαιότητα, μια ασφάλεια δικαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να επαναλάβω πως ο χρόνος ομιλίας είναι δύο λεπτά το πολύ για να μιλήσουν όλοι όσοι ζήτησαν το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γκρέτς από την Βουλή της Μάλτας. Σας ευχαριστώ. Οπωσδήποτε πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό και από πολιτική σκοπιά. Η σημασία και η ευαισθησία του συστήματος αυτού και η σημαντικότητά του άλλωστε απαιτούν ε, προσεκτική ανάλυση των συγκεκριμένων αυτών μέτρων στο κάθε κράτος μέλος. Συμφωνούμε με την δίκαιη φορολογία και είμαστε υπέρ πολλών ε, σημείων του πακέτου για την ε, φοροαποφυγή. Όμως δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα επηρεάζεται η κυριαρχία των κρατών μελών. Η φορολογία παραμένει εθνική αρμοδιότητα, γι' αυτό θεωρούμε πως έχει ζωτική σημασία εάν είναι να επιτύχει αυτή η πρωτοβουλία η επιτυχία αυτή θα έρθει πρώτα απ' όλα με το να σεβαστούμε πλήρως την αρχή της επικουρικότητας. όπως εξάλλου ε, ισχύει για ζητήματα φορολογίας όπου υπάρχει η πλήρης κυριαρχία των κρατών μελών. Τέλος, θεωρούμε πως σε μικρές οικονομίες οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε μεγάλους κινδύνους, μεγαλύτερους από ό,τι τα μεγάλα κρατημέλη, πρέπει να δούμε και τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό στις ε, οικονομίες μας έτσι ώστε οι πολίτες μας ε, να έχουν μία εμπιστοσύνη και να είναι υπέρ αυτού του πακέτου για να επιτύχουμε τον στόχο μας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ζολή έχει τον λόγο για τους πράσινους. Yes, good morning. Ναι. Χαίρετε. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία έκθεση που συνέταξαν οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, που ζήτησαν μάλλον ε, να συνταχθεί, για το IKEA. Διαπιστώσαμε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει αποφύγει ένα δις φορολόγηση σε έξι χρόνια. Έχω τα στοιχεία για πολλές από τις χώρες σας. Για παράδειγμα, για το Βέλγιο, 7 εκατομμύρια για ένα χρόνιο, 3 εκατομμύρια για τη Δανία, 23 για τη Γερμανία, 36 για τη Γερμανία και το καθεξής. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω να εξετάσετε το θέμα της επιχείρησης αυτής στη χώρα σας, να ρωτήσετε το Υπουργείο Οικονομίας και να εξετάσετε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ε, είναι διαθέσιμη η έκθεση, μπορώ να τη στείλω στη γραμματεία και μπορώ να την διαβιβάσω σε όλους. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι οι νέοι κανόνες BEPS ε δεν θα αλλάξουν ε, ε, τις πρακτικές αυτές. Δεν θα υποχρεωθεί η ΙΚΕΑ να πληρώνει φόρους εκεί που δραστηριοποιείται. Εμείς λοιπόν στο Κοινοβούλιο με την έκθεση που θα εκπονήσουμε θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να φροντίσουμε να καλύψουμε και αυτές τις μορφές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που δεν καλύπτονται από τα BEPS. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σοπρέα από την Γερουσία της Ρουμανίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. μην στηρίζουμε το σχέδιο δράση ω προτεραιότητα για την καταπολέμηση τη φοροαποφυγής από τι μεγάλε επιχειρήσει. Δεν πιστεύω να υπάρχει έλλειψη συντονισμού και τυποποίησης ώστε να έχουμε υψηλότερη συμβατότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Οπότε το σχέδιο οδηγία για το CCCTB είναι θετικό σύμφωνα με το Κρεβουλίο μας και δεν μπορεί να μας βοηθήσει για την καταπολεμιστή φορά αποφυγής. Θεωρούμε ότι ο στόχος μας εδώ θα πρέπει είναι να είναι το να αρθούν κάποια εμπόδια στην ενιαία αγορά και θα πρέπει να δούμε περισσότερο κάποια στοιχεία που περιλαμβάνει αυτή η οδηγία CCTV, λαμβάνοντα υπόψη του συνομικού ε, κινδύνους που θα μπορούσαν να υπάρξουν για την Ρουμανία. Η μείωση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα μειονέκτημα γιατί η επίτευξη εδώ είναι υψηλότερη όταν έχουμε μια αξία περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, από τη στιγμή που δεν έχουμε ενιαίε προδιαγραφές θα μπορούσαμε να έχουμε διακρίσεις και αβεβαιότητε όσον αφορά τους προϋπολογισμούς, του εθνικού προπολογισμού Το δεύτερο ήμιση του 2016 θα συνεχίσουμε να αναθεωρούμε το διοικητικό, μάλλον το δημοσιονομικό φόρτο αυτή τη πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή, η κυρία Λουαζέ από την Γαλλική Βουλή. Λουβαζή διορθώνει η ομιλητρία. Λουβαζή λέγομαι. Η σχέση του κύκλου εργασιών και τη φορολόγηση των κερδών είναι ένα βασικό σημείο στο οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει και να παρενέβει η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών και οι πληροφορίε που έχουμε λάβει δείχνουν ότι η βελτιστοποίηση νυφολογική, το εύρο τη και η εντατικοποίηση αυτών των πρακτικών χρειάζεται να μα κάνει να δράσουμε γιατί οι επιπτώσει είναι τεράστιε. Η ισότιμη φορολόγηση αποτελεί νομίζω ένα κλειδί, ένα σημείο κλειδί για την επιτυχία τη Ευρώπη. Δεν γίνεται αφενό να ζητάμε από του συμπολίτε μα Ευρωπαίου να συμμετάσχουν στις ε, δημοσιονομικές προσπάθειες και αφετέρου εμείς οι ίδιοι να μην αντιδρούμε αποτελεσματικά και δραστικά σε σχέση με τις πολυεθνικές. Θα πρέπει να παρανεύουμε και σε άλλα θέματα όπως η προάσπιση των ευρωπαϊκών καινοτομιών και να καταγγείλουμε ακριβώς τις ε, περιπτώσεις όπου έχουμε κατάχρηση της πόσες θέσης. Η αυτονομία βεβαίως των της ε, φορολογίας φορικών αρχών ε, στι χώρε μέλη πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα διασφαλιστεί. όμω θα πρέπει να έχουμε ε, προϊόντα τα οποία θα μα βοηθούν να αυξήσουμε τη διαφάνεια. Γι' αυτό ακριβώ άκουσα και την ανάγκη ύπαρξη εταιρικών σχέσεων που ανέφεραν οι με κάποιε χώρε. Αυτή η ανάγκη εταιρικών σχέσεων νομίζω είναι καθοριστικό στοιχείο για την υλοποίηση τη θεματολογίου BEPS. Σήμερα λοιπόν, όταν έχουμε τόσε μεταβολέ, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ακριβώ ότι η βούληση των χωρών μελών είναι εξασφαλισμένη ώστε πραγματικά να υπάρξει ουσιώδης φορολογική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. The next speaker on the... Ευχαριστώ πολύ. Ο από το Κοινοβούλιο της Δανίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι συνάλφοι βουλευτές. Ας θυμηθούμε τι είναι το BEPS. Το θέμα δεν είναι μόνο το να πάρουμε έσοδα από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Στόχο έχει να διασφαλίσουμε ότι οι μεγάλες ε, εταιρείες θα φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο οι εθνικές εταιρείες με τις πολυεθνικές. Αφορά και τον ε, θεμητό ανταγωνισμό μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Άκουσα λοιπόν κάποιε δηλώσεις σήμερα που αφορούν ε, την ε, ενημέρωση παραδείγματο χάρη του της κοινή γνώμης. Ε, Εμεί έχουμε κάνει τέτοια ενημέρωση στη Δανία, είμαστε αρκετά προοδευτικοί, όχι μόνο επειδή ήμουν εγώ ο αρμόδιος υπουργό. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Είχαμε συζητήσει το ζήτημα της ε, φορολόγησης των επιχειρήσεων εδώ και χρόνια και βλέπουμε πως ε, βλέπουμε αμερικανικές πολυεθνικές ε, επιχειρήσεις να έρχονται και να λένε γιατί δεν, να μην έχουμε περισσότερη διαφάνεια στην Δανία από τις άλλες χώρες. Όταν επιτύχουμε κάτι τέτοιο λοιπόν πραγματικά υπάρχει ε, πρόοδος. Αν μπορούμε λοιπόν κάτι να κάνουμε από την πλευρά της Δανίας ε, του Κοινοβουλίου για να σας βοηθήσουμε, είμαστε στην διάθεσή σας. Ε, έχουμε λοιπόν μια ανοιχτή βάση δεδομένων στη Δανία, έτσι ώστε βλέπει ο καθένας κάθε εταιρεία πόσο φόρο πληρώνει, πόσο έχει πληρώσει τα τελευταία χρόνια και αυτό πραγματικά αποτελεί ενημέρωση του κοινού. Αν υπάρχει κάτι λοιπόν το οποίο μπορεί να γίνει, ας το κάνουμε και ας περάσει το ΜΠΕΒΣ σύντομα ως νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Στόλογιαν από το ΕΛΚ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ε, ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε την ε, προσπάθεια αυτή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περάσει μια και να σταματήσει την ε, μετατόπιση των κερδών. Λέει γεγονός είναι πως οι μικρές και οι μισές επιχειρήσεις πληρώνουν περισσότερους φόρους από τις πολυεθνικές. Και πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική. Και μάλιστα μάθαμε από δηλώσεις κομισιών και Κοινοβουλίου πως ε, κάποιες από αυτές τις φορολογικές συμφωνίες παραβίαζαν τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και το ερώτημά μου προς Κομισιόν είναι πως ήταν δυνατόν να μην κάνετε τίποτα για αυτό το ζήτημα γιατί οι συμφωνίες αυτές υπάρχουν εδώ και χρόνια όχι ένα χρόνο ή κάτι μήνες και δεν κάναμε τίποτα. Και μόνο όταν έσκασε το σκάνδαλο δημοσίως κάνατε κάτι, όταν υπήρξε κατακραυγή. Αυτό είναι απαράδεκτο για Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Πώς μπορέσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο ή μάλλον να μην κάνουμε τίποτα εδώ και τόσο καιρό για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λόρη από το Κοινοβούλιο της Εστονίας. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τον Δανό συνάδελφο. Η καταπολόμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής είναι ο πρωταρχικός στόχος ε, της φορολόγηση των επιχειρήσεων και αυτό γιατί είναι θέματα θεμητού ανταγωνισμού και ο θεμητός ανταγωνισμός οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη και αυτό αναζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ και με αυτούς που επισημαίνουν ότι οι σημερινές οικονομίες δεν είναι αυτές που είχαμε στο παρελθόν. Τα φορολογικά συστήματα είναι παροχημένα. Παραδείγματος χάρη, η ψηφιακή οικονομία πολύ δύσκολα μπορεί να μας επιτρέψει να καταλάβουμε πού δημιουργείται η αξία. Αλλά θα πρέπει η φορολόγηση να γίνεται στο χώρο στον οποίο δημιουργείται το κέρδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καθορίσουμε πού υπάρχουν τα εισοδήματα και εκεί που δημιουργείται το εισόδημα, εκεί θα πρέπει να γίνεται και η φορολόγηση, στην πηγή. Το θέμα της εναρμόνισης των φορολογικών πληροφοριών και η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών θα πρέπει να έχει ως στόχο να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα διπλό ε, γραφειοκρατικό άχθος. Ε, χρειάζονται κίνητρα ε, όπως αυτά του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς προτείνουμε να το μετατοπίσουμε από το κεφάλαιο και την εργασία προς τους πόρους ε, και τη ρήπανση και αυτό θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα ανάπτυξη στην Ευρώπη. Κυρία Ανδρέα από, το, ε, από τη Γαλλική Γερουσία, ευχαριστώ. Το σχέδιο BEPS, ε το είπαν και οι συνάδελφοι, υποστηρίζεται ακράδαντα από τη Γαλλία. Το αναλύσαμε καταρχάς ε, στα πλαίσια της καταπολέμησης της ε, φορολογικής βελτιστοποίησης ε, και των μεγάλων ψηφιακών κολοσσών των ΗΠΑ. Πολλές όμως μεγάλες γαλλικές πολυεθνικές ανησύχησαν από την κατεύθυνση που παίρνουν στα BEPS και ο ρόλος της φορολογικής βάσης βοηθά αναδυόμενες χώρες όπως για παράδειγμα η Βρασιλία και η Κίνα να ε, βοηθήσουν ε, στη φορολογία μεγάλες γαλλικές πολυεθνικές. Ε, η φορολόγηση θα πρέπει να γίνεται στη χώρα στην οποία πολλούνται τα προϊόντα και όχι στη χώρα καταγωγής όπου υπάρχουν απλώς οι γενικές διευθύνσεις και έχουμε και τα πνευματικά δικαιώματα. Ε, στο Γερουσία, στη Γαλλία, διοργανώθηκαν μια σειρά από ακροασει προκειμένου να μπορέσουμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα της Γαλλίας να προασπίσει τα, επιχειρη... τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της ε, μέσω μιας φορολογικής διπλωματίας και στον ΩΣΑ αλλά και στα πλαίσια της ε, αναδιαπραγμάτευσης των φορολογικών συμφωνιών που επιβάλλονται. Ακούσαμε την ΩΣΑ, την δική μας φορολογική διοίκηση εγκρίθηκε από τη γερουσία συγκεκριμένη νομοθεσία. Έχουμε μεταφέρει κάποια από τα κριτήρια των BEPS, αλλά μας περιμένει πολλή δουλειά ακόμα και πρέπει όλοι να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής στον κατάλογο, ο κύριος Δεμάση από την ΚΟΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. welcome ορίζω στους αδέλφους της αυτά τα μέτρα πολέμηση είναι ένα μεγάλο βήμα και προς τη βοήθεια των πολιτών που υπεφέρουν ακριβώς από την δημοσίων πόρων νομίζω ότι αποτελούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις μια ενιαία οντότητα που πραγματικά είναι για τους κανόνες τώρα η Κομισιόν επέλεξε το επίπεδο εργαλείων του ΩΣΑ. Οπότε έχουμε εδώ το 30% όσον αφορά του τα, τα κέρδη προφόρων και την μεταφορά και τον έλεγχο των πολυεθνικών μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μεταφορά κέρδων. Όμως με το 40% κάτω από το επίπεδο των κανόνων CFC για τις μητρικές και το δραστή φορολογία, είχαμε αρχικά πρόταση 75, οι πανεπιστημιακοί είπαν 90%. Οπότε υπάρχει λοιπόν τεράστιο κίνητρο για την μεταφορά αυτών των επιχειρήσεων σε φορολογικού παραδείσους. Υπάρχει λοιπόν πολύ δουλειά ακόμα που θα πρέπει να κάνουμε και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μα εδώ στο Κοινοβούλιο ακριβώς για να πετύχουμε την φορολογική δικαιοσύνη, αυτό που χρειάζονται τώρα οι πολίτε μας και η ίδια η οικονομία, ώστε να χρηματοδοτήσουν τις δημόσιες επενδύσεις, να αποφύγουμε την, τις δραστηριότητα δραστηριότητας και να με το μελώνει αισιόδοξη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι για το θέμα του BEPS έχουμε δύο ερωτήσεις. Μία από την Βουλική Βουλή και μία από την Ρουμανική Βουλή. Να δώσω το λόγο και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια σύντομη απάντηση, δύο λεπτά ίσως και μετά να σας παραπέψω τι διμερείς συναντήσεις που μπορεί να έχετε εκτός αυτής της αίθουσας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, με χαρά να σας πω δύο λόγια για κάποια σημεία. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους αυτούς που αναφέρθηκαν στην απαραίτητη πορεία και ενοποίηση όλο αυτό που κάνουμε για τη μετατόπιση των μεγάλων επιχειρήσεων. Όλα αυτά στα πλαίσια του BEPS είναι απαραίτητα. Αλλά βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει μια εδρεωμένη στάση σχέση με την νέα αγορά. Δεύτερον, να μην σχολιάσω τις κρατικές επιδοτήσεις γιατί αυτό δεν αφορά την πολιτική της Κομισιόν. Δεν είναι και ο φάκελος με το οποίο ασχολούμαι. Αυτό το κάνουν αλφή του ανταγωνισμού. Να πω όμως ότι το θέμα της αναδρομικότητας που αναφέρθηκε δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο τις ε, μη συμβατές κρατικές επιδοτήσεις όταν αυτές ίσονται τέλος πάντων μη συμβατές και αποζημιώνονται. Να πω επίσης ε, και δύο λόγια για το βελγικό καθεστώς, για τους ονομαστικούς τόκους, ονομαστικά επιτόκια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε με κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή έχουμε συγκρίσιμα συστήματα σε άλλες χώρες μέλη, τα οποία συνδέονται από μέτρα αντικατάχρησης με μέτρα πολύ πιο αποτελεσματικά από αυτά τα, του Βελγίου. Αυτό είδαμε ας πούμε και αυτό υποβάλαμε στις στάσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμένου για το Βελγίο. Έχουμε ένα διάλογο επ' αυτού με το Βελγίο. Δεν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι απορριπτή από μόνο του, αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί βεβαίω με πολύ αυστηρούς κανόνες που καταπολεμούν τις καταχρήσεις όπως ας πούμε το Ιταλικό σύστημα το οποίο από αυτή την άποψη μας φαίνεται έτσι πιο εύρωστο από αυτό που ισχύει στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή. Αλλά ξαναλέω αυτό συζητιέται αυτή τη στιγμή με την πολιτική βελγική τάξη. Τώρα για το tax ruling της φορολογικές αποφάσεις να πω δύο πράγματα. Δεν ξυπνήσαμε μόνο μετά τις λουξοδιαρροές στην Κομισιόν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν. Αυτό το θέμα το συζητούσαμε εδώ και καιρό, το εξετάζαμε από το 2010. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα ήθελα να στηρίξω και να συμφωνήσω με τις θέσεις του συναδέλφου από τις κάτω χώρες ότι δηλαδή όταν έχουμε μια σωστή και φιλόδοξη νόμιμη βάση είναι πιο εύκολο να έχουμε θετικά αποτελέσματα από τι περιπτώσει όπου έχουμε κάποιε ρήτρε, οι οποίε επαφίονται στην καλή θέληση των χωρών μελών. Σήμερα λοιπόν έχουμε λοιπόν την οδηγία που αφορά τι φορολογικέ αποφάσει και είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι ώστε να διασφαλίσουμε ακριβώ την διαφάνεια από ό,τι ε, σε σχέση με το παρελθόν. Πάντω είμαι στην έθεσή σα για διμερή κουβεντούλα λόγω ακριβώ του περιορισμού χρόνου που έχουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και του άλλου ομιλητέ. Τελείωσε εδώ αυτό το μέρος συνεδρίασης. Περνάμε στο επόμενο μέρος για την Τραπεζική Ένωση. Να προσκαλέσω τον κύριο Φανρόη, τον συμπρόεδρο. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ. Okay. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, Εγώ και η συνάδελφος ε, από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να κάνουμε αυτές τις ε, ε, συζητήσεις και τώρα θα μιλήσουμε για την Τραπεζική Ένωση. Η Τραπεζική Ένωση είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη σταθερότητα του οικονομικού συστήματος στόχος αυτής της ε, ε, συνεδρίασης είναι να συζητήσουμε τι έχουμε επιτύχει μέχρι τούδε και καθώς επίσης και τις μελλοντικές προκλήσεις και να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε περαιτέρω την ε, Τραπεζική Ένωση. Ο νέος μηχανισμός επίλυσης διαφορών ε, είναι πλέον σε εφαρμογή και ε, καλωσορίζουμε σήμερα τους εκπροσώπους ε, των πρώτων δύο πυλώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Νουή, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον κύριο Κένι που είναι πρόεδρος του Single Resolution Board και θα ακούσουμε την εμπειρία τους για τους νέους αυτούς φορείς και τις προτεραιότητες για τις μελλοντικές τους εργασίες η, η σημερινή συνεδρίαση έρχεται μια μέρα μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Οίκων για την πρώτη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τραπεζική Ένωση, για την οποία εισηγητής είναι ο κύριος Γκουαλτιέρη. Στην έκθεση αυτή ε, κάνει έναν απολογισμό των εξελίξεων για την Τραπεζική Ένωση το 2015 και επιπλέον οι εργασίες στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης ε, καταθέσεων, το EDIS, έχει ξεκινήσει. Στην Ολλανδική Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπήρχαν ε, διάφορες απόψεις για την ανάγκη να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων αυτή τη στιγμή. Επομένως, ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η συζήτηση για την ολοκλήρωση του τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης. Προσβλέπουμε λοιπόν στην ανταλλαγή απόψεων ε, για την φιλοδοξία αυτή να υλοποιήσουμε τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταθέσεων σε μια αποτελεσματική τραπεζική ένωση ε, και έτσι να σταματήσει η σχέση μεταξύ κυριαρχίας και τραπεζών, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών και να διασφαλίσουμε οικονομική σταθερότητα. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Ντανιέλ Νουή, πρόεδρο του ε, Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ευχαρίστηση κυρίες και κύριοι βουλευτές το ότι βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα σε αυτή την ε, συνεδρίαση της ε, Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής. Είχα προγραμματίσει να σας μιλήσω για δύο ζητήματα. Πρώτα, ποια είναι τα επιτέγματα του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού το πρώτο έτος και δεύτερον, σε ποιο βαθμό εμποδίζουν την αποτελεσματική εποπτεία οι διαφορετικοί εθνικοί τραπεζικοί κανόνες. Όμως δεδομένη τη κατάσταση στις αγορές νομίζω πως λογικότερο είναι να σα πω πρώτα απ' όλα ποια είναι η αξιολόγησή μας για την κατάσταση στον τραπεζικό τομέα αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας πως η κατάσταση σήμερα είναι πάρα πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν το 2012. Ο τραπεζικός τομέας είναι πολύ πιο ανθεκτικός καθώς ο λόγος ε, των ε, κεφαλαίων ε, Tier 1 είναι, ε, έχει αυξηθεί από 9% 2012 σε 13% περίπου μετά την δική μας διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης, το λεγόμενο SREP. Επιπλέον η ποιότητα του κεφαλαίου των τραπεζών έχει βελτιωθεί σημαντικά, άρα ο κλάδος είναι, έχει την ικανότητα να απορροφήσει αναπάντηχες εξελίξεις πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Υπάρχουν βεβαίω ακόμα κάποιε τράπεζε που έχουν υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όμω, κατά τη διάρκεια τη συνολική αξιολόγηση, τα δάνεια αυτά τα έχουμε ταυτοποιήσει χρησιμοποιώντα για πρώτη φορά έναν κοινό ορισμό που μα έδωσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ταυτόχρονα. Έχουν γίνει και επαρκεί προβλέψει για τα μη εξυπηρετούμενα αυτά δάνεια. Οπότε είμαστε σε μια λογικά άνετη θέση για να συνεχίσουμε να μειώνουμε αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με έναν τακτικό τρόπο τα επόμενα χρόνια. Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές έτσι ώστε να συμπληρώνται τα δικά μας τα μέτρα με τα απαραίτητα εθνικά μέτρα. Με τον κύκλο λοιπόν ΣΡΕΠ της αξιολόγησης του 2015 τονίσαμε τις ε, απαιτήσει ε, τις κεφαλαϊκές του πυλώνα 2 που αναμένουμε να δούμε στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό σημαίνει πως αν δεν αλλάξουν τα πράγματα οι κεφαλαϊκές απαιτήσει δεν θα αυξηθούν άλλο. Οι σημαντικές ε, τράπεζες υπό την υποπτία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις της, σχετική της σχετικής 4 μέχρι το 2019. Μάλιστα οι περισσότερε από αυτές το έχουν ήδη καταφέρει και οι υπόλοιπε αντιμετωπίζουν μια σταδιακή εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών και έχουν πολιτικές κατανομής των κερδών οι οποίες θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν τις νέες απαιτήσεις μέχρι την προθεσμία του 2019. Το 2015 οι τράπεζες υπό την υποπτία της ΕΚΤ άξαν περτέρω τα κέρδη τους σε σχέση με το 2014 και έτσι μπορούν να έχουν την κατάλληλη πολιτική διανομής ε, κερδών ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνονται, ανταποκρίνονται στις νομικές ε, απαιτήσεις κεφαλαϊκής επάρκειας δανείζοντας ε, και στην οικονομία. Επίσης ο κλάδος έχει αποθεματικά για να ανταποκριθεί στα κεφαλαϊκά μέσα Tier 1 και βεβαίως ε, καθώς έχουμε σταδιακή εισαγωγή των απαιτήσεων αυτών οι τράπεζες ήδη υπερβαίνουν τα ελάχιστα κατόφλια και συνεχίζουν να σχηματίζουν αποθεματικά. Έχουμε λοιπόν τώρα μία οδηγία την BRD η οποία είναι οδηγία διάσωσης ε, και αναδιάρθρωσης ε, τραπεζών στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Ενώ λοιπόν αυξάνεται η πειθαρχία της αγοράς για επενδυτές και τράπεζες, η πρόσφατη αύξηση στις ψαλίδες ε, δεν μας φαίνεται δικαιολογημένη δεδομένου των πολύ υψηλότερων ε, επιπέδων κεφαλαίου που έχουν οι τράπεζες που είναι πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσει. Αυτά τα πράγματα για την τωρινή συγκυρία. Τώρα θα ήθελα να αφαιρθώ στα σημεία για τα οποία με είχατε αρκετά καλέσει. Πρώτα απ' όλα για αυτά τα οποία πέτυχε ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός το πρώτο έτος. Εφόσον πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο τραπεζικός επόπτης για ολόκληρη την Ευρωζώνη και δεδομένου του ελάχιστου χρόνου που είχαμε στην διάθεσή μας, θεωρώ πως αυτό ήταν ένα επίτευγμα. Και βεβαίως ε, βασικό κομμάτι της προσέγγισης μας είναι να αντιμετωπίζουμε όλες τις υποπτευόμενες τράπεζες με τα ίδια χαρακτηριστικά με τον ίδιο τρόπο. Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειαζόταν δύο πράγματα. Ενιαίους ε, κανόνες και ενιαίο τρόπο εφαρμογής. Από όταν λοιπόν ε, συστάθηκε ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και έχουμε τώρα μια κοινή μεθοδολογία όσον αφορά την ε, εποπτική αναθεώρηση και τη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει πως έχουμε αυστηρές και δικές εποπτικές απαιτήσει και πηγαίνουμε προς ίσους όρους ανταγωνισμού στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Όμως δεν έχουμε ενιαίους κανόνες αυτή τη στιγμή, οπότε η πλήρης εναρμόνιση δεν είναι ακόμα δυνατή. Ένα ζήτημα εδώ πέρα είναι οι λεγόμενες επιλογές και η διακριτική ευχέρεια που υπάρχει στο εθνικό επίπεδο. Κάποιες από αυτές τις επιλογές βεβαίως είναι επιλογές που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μπορώ να σας πω πως θα περάσουμε σε μια εναρμόνιση για τις περισσότερες από αυτές κατά τη διάρκεια του 2016, οπότε το ερώτημα είναι το εάν οι διαφορετικοί εθνικοί κανόνες δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική και ενιαία υποπτία. Υπάρχει ένα όριο ότι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν διαφορές τις οποίες δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς και βεβαίως οι αποκλήσεις αυτές διαταράσσουν τους ισόρους ανταγωνισμού. Οι αποκλήσεις αυτές λοιπόν έχουν διάφορες αιτίες. Πρώτα απ' όλα η νομοθεσία της Ένωσης αυτή τη στιγμή δίνει επιλογές και στα κράτη-μέλη ε, για να περάσουν εθνικούς νόμους. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για περαιτέρω εναρμόνιση. Εδώ πέρα απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία για να διορθωθεί το πρόβλημα στην πηγή. Δεύτερον, μια σημαντική πηγή αποκλήσεων είναι ε, το ότι έχουμε οδηγίες αντί για κανονισμούς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τη στιγμή στην οποία απαιτείται γρήγορη παρέμβαση της ρυθμιστικής αρχής είναι όταν μια τράπεζα έχει προβλήματα. Γι' αυτό ακριβώς η οδηγία BRD έδωσε στον, στην εποπτική αρχή δυνατότητες έγκαιρης παρέμβασης. Όμως, μια που είναι οδηγία της ε, Ένωσης, η μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο ήταν υπόθεση των κρατών μελών. Ε, ως αποτέλεσμα αυτού, Έχουμε 19 διαφορετικά νομοθετήματα στην Ευρωζώνη. Η ενιαία νομοθεσία στον κλάδο αυτόν, ένας κανονισμός, είναι κάτι το οποίο είναι όχι απλά επιθυμητό, αλλά αναγκαίο. Τρίτον, η εθνική νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει επίσης πρόβλημα στους ίσους ανταγωνισμού στην Τραπεζική Ένωση, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ανάγκη να μεταφερθεί ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για εναρμόνιση των κανόνων περιορίζεται από τους επιπρόσθετους κανόνες που επιβάλλει το Εθνικό Δίκαιο κάποιων χωρών. Σε κάποιες χώρες, π.χ., μη δεσμευτικές εποπτικές πρακτικές μετατρέπονται σε δεσμευτικά νομοθετήματα. Για να επιτύχουμε μια πραγματική τραπεζική ένωση, τα κράτη-μέλη άρα θα πρέπει να μην ε, δημιουργούν φραγμούς σε ενιαίες εποπτικές πρακτικές και στην ε, διακριτική ευχέρεια που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή. Να καταλήξω λοιπόν, το ενιαίος εποπτικός μηχανισμός δημιουργήθηκε από τον κοινοτικό νομοθέτη με στόχο με ένα συγκεκριμένο στόχο και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον επιτύχουμε. Υπάρχουν όμως κάποια όρια και εδώ πέρα ακριβώς χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας ημών των ομοθετών και στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο για να επιτύχουμε μια πραγματικά ενιαία υποπτία. Πρέπει να συνεργαστούμε για να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό και πρέπει βεβαίως να είμαστε πάρα πολύ σε επιφυλακή και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι προληπτικοί κανόνες για τις τράπεζες να είναι πλήρω εναρμονισμένοι για να επιτύχουμε την αποστολή που μας έχετε αναθέσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νόη. Στον κύριο Κένιχ να δώσουμε τώρα το λόγο. Στην κυρία Κένιχ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Κοινοβουλίου. Επειδή είμαστε μια νέα οργάνωση στα πλαίσια του SME, Έχω την ευκαιρία για πρώτη φορά να μιλήσω ταυτόχρονα και σε εθνικούς αλλά και σε ευρωβουλευτές. Να σας πω ότι έχουμε μία δέσμευση για την διαφάνεια και χαίρομαι που έχω την κυρία Νουή δίπλα μου γιατί βλέπω ότι έχουμε πολλά να πούμε κοινά Κατευθείαν λοιπόν να πάω στα δύο ζητήματα που μας αφορούν επιτεύγματα του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού το 2015 και οι προτεραιότητες για το 2016. Και στο τέλος θα σχολιάσω το αρχικό σχολείο της Δανιέλ με το οποίο σφωνώ Είχαμε λοιπόν πολλά επιτεύγματα για το ΣΕΜΙ το 2015 Πήγα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ πριν από δύο εβδομάδε οπότε θα προσπαθήσω να αποφύγω αυτά που είπα εκεί, αλλά βεβαίω υπάρχει μια φράση που ξαναλέω, που λέω συνέχεια, ότι βρισκόμαστε στην αρχή. Έχουμε ένα προσωπικό τότε 30 υπαλλήλων, ελπίζουμε να διπλασιαστεί μέχρι το τέλο του τρέχοντο έτου Και οργανωνόμαστε και έστω και αν αρχή τα πράγματα πάνε καλά, αλλά βέβαια μπορούν ακόμα να γίνουν πολλά. Για το περιεχόμενο τώρα. Ήδη ήμασταν έτοιμοι από πέρσι, όπως αναφέρει και εκεί έκθεση του και πραγματικά προσπαθήσαμε σκληρά ώστε τους τελευταίους μήνες να είμαστε πλήρως έτοιμοι αναλαμβάνοντας ακριβώς δράσεις που αφορούν το αντικείμενό μας στις αρχές του τρέχοντος έτους. Είχαμε αρχικά διαπραγματεύσεις και οδήγησαν αυτές σε μια συμφωνία που υπογράφει τον Δεκέμβρη Λέχεια συμφωνή νωρίτερα μεταξύ του Κοινοβουλίου και του ΕΣΜΗ e όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ε, Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας και του ΕΣΜΗ e για ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία. Όλα αυτά ε, είναι ολοκληρωμένα και βεβαίω έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με ανταλλαγή στοιχείων τα οποία έχουν τεράστια σημασία και για μα. Εμεί είμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία βεβαίω με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για όλα αυτά τα θέματα και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ένα από αυτά τα ζητήματα που ζητάμε η Ντανιέλ και εγώ όλο και πιο συχνά όταν βρισκόμαστε. Η στενή λοιπόν συνεργασία θα πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι που ήδη έχει υλοποιηθεί με τις εθνικές αρχές και αυτό είναι βασικό επειδή οι εθνικές αρχές ε, εκαθάρισης νομίζω ότι διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα αλλά έχουμε και τους μηχανισμούς ε, μεταφοράς οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι η γνώση εθνική και τα εθνικά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά στις δράσει μας. Έχουμε συντάξει ή βρισκόμαστε ε, στα τελευταία στάδια σύνταξη ενό χειριδίου κρίσεως μαζί με τον ΡΑΕΣ και ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε μια σταθερή διαδικασία εκαθάρισης και αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε διαδικασίες εκαθάρισης στην ζώνη του ευρώ στο άμεσο μέλλον αποτελεσματικά. Και χάνει διαφάνειας προτιθέμεθα να δημοσιεύσουμε ένα σύντομο έγγραφο το οποίο θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές παράλληλα με το εποπτικό εχειρίδιο αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους ώστε όλος ο κλάδος αλλά και η κοινή γνώμη να, να καταλάβουν ακριβώς πώς σχεδιάζουμε το θέμα της εκαθάρισης και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να διασφαλίσουμε την ύπαρξη διαφανέ και ασφάλεια στι αγορέ. Η συνεργασία και ο συντονισμό με τι αρχές αρχέ, εκτό από τη συνεργασία και το συντονισμό με την ε, Κεντρική Τράπεζα, έχει τεράστια σημασία, αλλά δεν επαρκεί, οπότε θα πρέπει να συντονιστούμε και να συνεργαστούμε διεθνώ, εκτό δηλαδή ζώνη ευρώ και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι περισσότερες από τις μεγάλες τράπεζες ασκούν δραστηριότητε και εντό και εκτό ζώνη ευρώ. Νομίζω ότι θα ήταν σωστό να πούμε και συμφωνεί αυτό με αυτά που είπατε και εσεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά όχι μόνο στο θέμα τη εποπτεία αλλά και στα θέματα σχεδιασμού εκαθάρισης. Αλλά παραμένουν βεβαίω θέματα ακόμα ανοιχτά, γι' αυτό ακριβώ αναφέρθηκα, μάλλον είπα ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και τι πατριωτές μα για το 2016. Το αποτελεί έναν οργανισμό ο οποίος ε, κοιτάει στο μέλλον. Οπότε σχεδιάζουμε τα θέματα καθάρισης με την πεποίθηση ότι ο σωστός σχεδιασμός καθάρισης θα αποφύγει τις σοβαρές ε, επιπτώσεις των καθαρίσεων, οπότε ε, δεν περιμένουμε έτσι, τους πελάτες μας να χτυπήσουν την πόρτα μας, το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου αυτό. Κύριος στόχος μας για το 16 σε αυτόν τον τομέα, σχεδιασμός των καθαρίσεων, είναι το να έχουμε την ε, πλήρη δυνατότητα να χαράξουμε σχεδιασμό και σχέδια για τις εκαθαρίσεις για όλα για όλες τις οντότητες που βρίσκονται στο πεδίο αρμοδιότητές μας και με όλους τους εμπλεκόμενους. Και ένα πολύ σημαντικό τμήμα αυτής της διαδικασίας είναι βεβαίως το να καθορίσουμε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τα ίδια κεφάλαια, το περιβόητο εμπράλ, για όλες τις οντότητες και όλες τις ομάδες που μας αφορούν. Αυτό θα ολοκληρωθεί, ελπίζουμε, πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους και το ΕΜΡΑΛ θα αφορά όλες τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο σωστό και αναλογικό. Έργο μας θα είναι να ευθυγραμμίσουμε κάποιες από τις διεθνείς απαιτήσει, το TLEC, έτσι λέγεται, με το ΕΜΡΑΛ και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η προσέγγιση θα είναι σωστή και το καλό εδώ είναι ότι αυτό γίνεται, είναι εφικτό και αυτό το κατανοεί βεβαίως και ο χρηματοοικονομικός κλάδος. Το Emerald ε, αποτελείται από το ποσοστό αυτό το 8% των δύο κεφαλαίων, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ε, έχουμε να κάνουμε ψηλότερα ποσοστά για τις μεγάλες τράπεζες στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έμπρα δεν σημαίνει βεβαίω ότι θέτουμε ποσοτικά στοιχεία ή ποσοτικού στόχου ανά τράπεζα. Βεβαίω θα έχουμε ποσοτικού στόχου, αλλά δεν θα αποτελέσουν μοχλοποίηση προ αυτέ. Μετά θα πρέπει να αποφασίσουμε βεβαίω και για ποιοτικά στοιχεία, τα οποία ενδεχομένω θα είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστούν και μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο οι τράπεζε για να προσαρμοστούν σε αυτά, αλλά θα το κάνουμε περίπτωση ώστε πραγματικά οι τράπεζες στο μέλλον να είναι σε θέση να είναι σε εύρωστη οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε και όπως έλεγε και η Ντανιέλ προηγουμένως υπάρχει και ένας τομέας όπου χρειάζεται περισσότερη ενότητα από ποικιλομορφία δηλαδή η αξιολόγηση των, α, της πιστοτικής η BRD, ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται με νέο τρόπο, ώστε να έχουμε μεταφορά βεβαίως που τον Playbird, αλλά όχι, έχουμε μεταφορά τώρα, αλλά όχι με νέο τρόπο. Αυτό βεβαίω δεν είναι καταστροφικό, αλλά μα δυσχεραίνει. Οπότε σε κάποιε περιπτώσει αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ε, σε διαδικασίε λιγότερο ομαλέ ή λιγότερο θετικά αποτελέσματα. Να σας ε, ενημερώσω και για το νέο Ταμείο Καθάριση. Έχουμε τις ρυθμίσεις που αφορούν τα δάνεια, οι οποίες ε, συμφωνίε έχουν υπογραφεί και θα γίνουν περισσότερα τι επόμενε εβδομάδε. Έχουμε επίση συλλέξει και τις συνεισφορές για το 2015. Αυτό έγινε στα τέλη του Γενάρη. Μας μεταφέρθηκαν αυτές οι συνεισφορές. 4,3 δις είναι αυτά. Σύμφωνα δηλαδή με αυτό που αναμέναμε. Τώρα, για τις συνεισφορές του 16 θα μεταφέρουν στο SRF στις 30 του Ιούνιου και μετά θα έχουμε τα δύο χρόνια αυτά συνεισφορών που θα έρθουν εδώ. Και επειδή τελειώνει και ο χρόνος μου, να επανέλθω σε αυτό που είπε η Ντανιέλ προηγουμένω ότι θα μπορούσαμε να πούμε από το 2008-2009 έχουν γίνει πολλά είναι πιο εύρωστα οι τράπεζες έχουν λιγότερη μόχλευση είναι σε καλύτερη θέση ε, ακόμα και σε σχέση με, τη, με την κορυφή της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως Ένωση είμαστε πιο ανθεκτικοί στα οικονομικά ΣΕΚ και νομίζω η BRD μα ε, παρέχει σε περίπτωση που σημαίνει κάτι ένα πλαίσιο εκαθάρισης. Δεν έχει γίνει από το 2014 αυτό βέβαια και γι' αυτό ακριβώς είμαστε δεσμευμένοι στο να τα αφαρμόσουμε αυτά με τρόπο διαφανή και σταθερό. Νομίζω η έννοια της ε, περιπλοκότητας στην Ευρώπη είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά όσον αφορά τις εκαθαρίσεις νομίζω το BRD μας ε, παρέχει ακριβώς σαφείς ε, κατευθύνσεις για το καταμερισμό των βαρών και ελπίζουμε από τον οργανισμό μας να τα πετύχουμε όλα αυτά με τρόπο σωστό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρομπέρτο Γουαλτιέρη, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και εισηγητή για την πρώτη ετήσια έκθεση για την ε, Τραπεζική Ένωση. Παρακαλώ κύριε Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Πράγματι είναι χαρά να βλέπω εδώ τους δύο βραχίονες της Τραπεζικής Ένωσης μαζί. Το ε, Κοινοβούλιο ήταν ένθερμος υποστηρικτής αυτού του προ, του σχεδίου. Επομένως θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονός ότι στην πρώτη μας έκθεση, η οποία εγκρίθηκε μόλις εχθές ε, με μεγάλη πλειοψηφία, 71% της Επιτροπής, επομένως έχουμε μια γενική αξιολόγηση αυτή της πρώτης χρονιάς της Τραπεζικής Ένωσης, κυρίως ε, το SSM και το πρώτο βήμα του SRM, ε, του Ενίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, που είναι ένα θετικό βήμα. Το Κοινοβούλιο λοιπόν σύσσωμο πιστεύει ότι η σύσταση του SSM ήταν επιτυχία και από επιχειρησιακή σκοπιά και από πλευράς ε, ε, ποιότητας της εποπτείας. Από επιχειρησιακή σκοπιάς ε, θεωρούμε πράγματι αξιοσημείωτα τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι τούδε, ιδίως σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και βεβαίως ε, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την ποιότητα της ε, συνεργασίας με τους εποπτικούς φορείς και ε, σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο μπορούμε επίσης να εξορθολογήσουμε και κάποιες ε, διοικητικές διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όσον αφορά την πολιτική εποπτείας, πιστεύω πράγματι ότι το Εποπτικό Συμβούλιο έχει συνεισφέρει ιδιαίτερα το SSM για την αποκατάσταση της ε, ε, δύναμης και της ανθεκτικότητας του τραπεζικού μας συστήματος. Ε, συμφωνώ και με αυτά που μόλις είπε η κυρία Κέννη και συμφωνώ με την άποψή της για τη βελτίωση στην ποιότητα και την ποσότητα των δυνατοτήτων που διαθέτουμε. και μάλιστα κάποιες από τι πρόσφατε εξελίξεις στην αγορά δεν αντικατόπτριζαν ε, κάποια πράγματα. Υπάρχουν διάφορα δεδομένα που μπορούμε να διαβάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και ε, ένας από τους παράγοντε που συνεισφέρει στο θέμα αυτό είναι και η ποιότητα τη ε, δράσης εποπτείας σε αυτή την πρώτη χρονιά. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες παρατηρήσεις κυρίως για ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με το λεγόμενο MDA, το Minimal Distributable Amount, που είναι ε, ένα στοιχείο το οποίο δεν θεωρούμε ότι είναι αρκετά σαφές στην παρούσια νομοθεσία, αλλά θα μπορούσαμε ίσως εδώ να χρησιμοποιήσουμε κάποια μεγαλύτερη ευελιξία για να δούμε τι γίνεται με τις 81 αγορές ομολόγων. Δεν ξέρω αν ε, ε, γνωρίζει και η Ντανιέλ ε, αν εν ώψη και αυτή τη πρόσφατη εξέλιξη θα μπορούσαν να εξετα... επανεξετάσουν την προηγούμενη απόφαση για να χρησιμοποιήσουν πλήρω την ευελιξία που κατά την άποψή μα μπορεί να υπάρξει. Μετά υπάρχει και το θέμα της αναθεώρησης της νομοθεσίας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα, ε, παραδείγματος χάρη το, να έχουμε στο ίδιο καλάθι ομόλογα θέματα του 81 και το καθεξής. Υποστηρίζουμε βέβαια και οποιαδήποτε προσπάθεια σε νομοθετικό επίπεδο, υποστηρίζουμε και την ε, προαιρετική διακριτική ευχέρεια της κάθε χώρας. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουν τεθεί σε διαβέουλευση στον τομέα αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές υποστηρίζουμε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια, όπως επίσης πρέπει να πω υποστηρίζουμε και μια γενικότερη συμφωνία για μια, για μια νομοθετική παρένθεση. Πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα αναγνωριστεί και κάπου που δεν το περιμένετε. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αναγνωρίζεται ότι ε, ένα περαιτέρω επίπεδο εναρμόνισης θα έπρεπε να υπάρχει στην Τραπεζική Ένωση. Υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο ισχύει για όλους και είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει και ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου ότι θα παραμείνει. Και υπάρχει λοιπόν ένας ενιαίος οδηγός ε, και επίσης χρειαζόμαστε και περισσότερα συγκεκριμένα μέτρα για την εναρμόνιση που είναι χρήσιμα και σημαντικά και συμφωνώ και τα υποστηρίζουμε όλα αυτά. Υπάρχει και το θέμα της δυνατότητας να αξιολογήσουμε την εποπτεία των τραπεζών, τα ισοζύγια τους, τις τραπεζικές τους δραστηριότητες. Πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε πέραν του επιστοτικού κινδύνου και να δούμε όλες τις μορφές ε, τραπεζικού κινδύνου, παραδείγματο χάρη ε, τα χρηματοπιστωτικά χαρτοφυλάκια και ε, εισοδήματα κατηγορίας 3, στοιχεία μάλλον ενεργητικού κατηγορίας 3. Υπάρχει επίσης και το SRM, το Ενίο Συμβούλιο Εξυγίασης, το οποίο όπως είπε και η κυρία Κόνικ είναι ακόμα στην ε, αρχή του, αλλά εμείς ε, τα υποστηρίζουμε όλα, υποστηρίζουμε και την αρχή του Μπέιλιν, τη διάθεση με ίδιου πόρου. θεωρούμε ότι είναι μια σωστή αρχή και δεν θα πρέπει να χαθεί αυτή η βασική αρχή. Γίνεται μεγάλη συζήτηση σε κάποια κράτη-μέλη ε, αυτό σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στην νομοθεσία και να αξιολογήσουμε προσεκτικά τις διάφορες επιλογές που είναι στη διάθεση του Συμβουλίου με βάση την τρέχουσα νομοθεσία, καθώς επίσης και διάφορους τρόπους ε, εξυγίανσης πέραν της εκαθάρισης και φυσικά κατάλληλη αναλογικότητα, δικαιοσύνη, ευελιξία, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο νομοθετικό πλαίσιο. Και φυσικά όλα αυτά μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια αφενός, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να διαφυλάξουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα ΦΕΤΕΛ. Και τέλο υπάρχει το θέμα της ολοκλήρωσης τη Τραπεζική Ένωση. Ε, πιστεύω ότι είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ε, καλωσορίζει τη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Θα δούμε βέβαια και το περιεχόμενο. Το Κοινοβούλιο θα ακολουθεί στη δέουσα νομοθετική διαδικασία, δεν προβλέπουμε κάποια συγκεκριμένη αξιολόγηση, αλλά είμαστε θετικά διακείμενοι σε αυτή την αξιολόγηση και φυσικά ε, υποστηρίζουμε τα πράγματα αυτά με κάποια επιφύλαξη βέβαια ε, για το συγκεκριμένο τομέα της ε, κυρίαρχης θέσης των κρατών μελών. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μια συμβιβαστική διατύπωση και θα πρέπει να γίνει μεσοπρόθεσμα στα πλαίσια των διεθνών φορέων και την Επιτροπή ε, Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και φυσικά να αποφύγουμε και ε, συγκεκριμένες συνέπειες για την αγορά, κυρίως ακούσιες. Εχθέ ο κύριο Δράγκη μα εξέφρασε και τι απόψει του και πρέπει να πω ότι συμφωνώ απολύτω ε, με την άποψή του. Αυτά λοιπόν σε γενικέ γραμμέ για την άποψή μα και ε, θα ήθελα να επισημάνω λοιπόν αυτά τα σημεία τα οποία σας επισήμανα και φυσικά ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε περαιτέρω και με το Συμβούλιο Εποπτείας ε, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με το Νέο Συμβούλιο Εξυγίανση και να δούμε πώ μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή την Τραπεζική Ένωση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην ε, κυρία Χιούμπνερ. Πού είναι? Α, εκεί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής είναι σαφές νομίζω πως η Τραπεζική Ένωση είναι ακόμα ανεξελίξη. Κοίτοντας το μέλλον λοιπόν, καλό είναι να θυμόμαστε πως ε, ξεκίνησε η Τραπεζική Ένωση για να σπάσει ε, ο δεσμός μεταξύ τραπεζών ε, και κρατών για να μην πέφτουν οι τράπεζες στα προβλήματα του δημοσίου χρέους και βεβαίως να μην ξεχνάμε και τις διάφορες εξωτερικότητες και ότι δεν μπορεί να υπάρχει αποτελεσματική εποπτεία μεγάλων διασυνοριακών τραπεζών. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και να θυμόμαστε γιατί ξεκινήσαμε και η γνώση είναι πως ε, πολλά έγιναν και η παρουσίαση και των κύριων ε, Λουί και Κένιγκ μας έδωσε τα σχετικά στοιχεία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα ξεκινάμε την εργασία σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων κατά το οποίο βέβαια είναι μια σταδιακή διαδικασία αλλά ως συνήθως όσο πιο πολύ ολοκληρώνουμε μια ομάδα, ένα πυρήνα καρτών, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση μια Ευρώπη σε δύο ταχυτήτων και υπάρχουν αποκλήσει μεταξύ αυτών που είναι μέσα και εκτός. Και ακριβώς θα πρέπει να διατηρήσουμε το σύστημα ανοιχτό για τις χώρες εκτός ευρωζώνη, δηλαδή να κάνουν κάποια συμφωνία συνεργασία με τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό και έτσι αυτομάτως θα είναι και στο πλαίσιο του ενιαίου μηχανισμού διάσωσης. Βεβαίως γεγονός είναι πως ε, η καμία κυβέρνηση δεν έχει ακόμα εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αν και πέρσι η κυβέρνηση της Δανίας ε, είπε πως θα ήταν προς το συμφέρον της. Η Δε Σουηδία είπε πως δεν θα ήθελε να ενταχθεί. Έχει κάποια θετικά αυτή η προσέγγιση του βλέποντας και κάνοντας, αλλά τελικά είναι προς το συμφέρον αυτών των χωρών να ενταχθούν. Η Τραπεζική Ένωση είναι κάτι το οποίο εμβαθύνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είναι ανοιχτό, όπως είπα, σε όλους. Όλοι μπορούν να ενταχθούν εάν θέλουν και αλλιώς θα μείνουν έξω και θα υπάρχει ο κίνδυνος περιφερειοποίησης. Συχνά το θέμα είναι πως οι χώρες οι οποίες είναι εκτός ευρωζώνης είναι αυτές ακριβώς οι οποίες χρειάζονται μια πανευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα αυτό της ε, διάσωσης. Και βεβαίως ε, βλέπουμε πως ε, μεγάλο κομμάτι σχεδόν ενεργητικού το έχουν στην κατοχή τους ξένες ε, τράπεζες και διασυνοριακοί όμιλοι ακριβώς ε, αυτά τα χρηματοπιστωτικά εντρήματα των οποίων η υποπτία είναι ιδιαίτερη δύσκολη και για τα οποία έχει σχεδιαστεί η Τραπεζική Ένωση επιπλέον τα στοιχεία αυτά τα οποία κατέχουν οι ξένες τράπεζες δεν τα έχουν τράπεζες τρίτων χωρών αλλά κυρίως τράπεζες με έδρα εντός Τραπεζικής Ένωσης. Π.χ. στην Τσεχία υπολογίζεται πως 88% των διαφόρων στοιχείων ενεργητικού είναι στην κατοχή διασυνοριακών τραπεζών ε, και κυρίως μιλάμε για τράπεζες της ε, περιοχής της Τραπεζικής Ένωσης, τα ίδια και στη Βουλγαρία. Να πω λοιπόν πως ε, καλό είναι οι χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη και σκοπεύουν να μπουν να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην Τραπεζική Ένωση. Σας ευχαριστώ κυρία Χίμπνερ. Η κυρία Κάριν Μπερζιέ έχει τώρα τον λόγο. Από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, μέλος τη Επιτροπής Οικονομικών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρητήρια καταρχάς στην κυρία Νοή και στην κυρία Κένικ για τη δουλειά τους. Έχει απόσταση το να πρέπει να αποφάσισουμε να εφαρμόσουμε. Τρία σημεία σύντομα. Καταρχάς, τι γίνεται με τη Γαλλία όσον αφορά την εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης. Έχουμε προχωρήσει για αυτό το θέμα και όσον αφορά τους μηχανισμούς εξυγίανσης η Γαλλία έχει λάβει απόφαση ήδη από το 2013 και για το σύνολο των μηχανισμών εποπτείας όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Τραπεζική Ένωση ήδη έχουν εφαρμοστεί στη Γαλλία. Από αυτή λοιπόν την άποψη και για το θέμα στο οποίο θα επανέλθω των τραπεζικών εγγύσεων η Γαλλία ως χώρα α, μέλος ήδη έχει προχωρήσει λοιπόν. Οπότε η Γαλλία όχι μόνο στηρίζει αυτή την εξέλιξη αλλά κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να εφαρμόσουμε και να ανταποκριθούμε σε αιτήματα που αφορούν τις διάφορες, ε, και σχετίζονται με τις διάφορες οδηγίες της, οδηγίες της Ένωσης. Μετά, να μιλήσω τώρα για το διακύβευμα της μελλοντική Τραπεζικής Ένωσης. Όντως έχουμε κάνει πολλά. Όντως μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την περισσότερη ολοκλήρωση όσον αφορά τον έλεγχο του, χρωμα, οικονομικού τομέα με τους δύο πυλώνες, δηλαδή εποπτεία και εξυγένση. Ενιαία εποπτεία και εξυγένση, ενιαία λοιπόν εποπτεία και εξυγένση αποτελούν σημαντικές πρόοδους και αν μια μέρα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους μηχανισμούς πανευρωπαϊκά δεν θα το πιστέψουν και πολύ. Χαιρόμαστε λοιπόν που υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά συγκεκριμένα για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Η συζήτηση σήμερα μας δείχνει ότι είμαστε ακόμα σε πολύ τεχνικό και αφηρημένο και μακροοικονομικό επίπεδο. Για τους πολίτες λοιπόν και τις πολίτησε της Ευρώπης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλιστεί την μέρα που τα δικά σου τα χρήματα θα είναι εγγυημένα, που οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι εγγυημένες, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε εμπιστοσύνη και θα προστατευτούν όλα αυτά από το σύνολο των μηχανισμών που έχουμε δημιουργήσει. Η Τραπεζική Ένωση διέρχεται ακριβώς από την οικοδόμηση της Ευρώπης, την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οπότε πρέπει να πάμε μέχρι το τέλος. Δηλαδή θα πρέπει να καταλήξουμε στην εγγύηση των καταθέσεων που όπως είδαμε με την Κυπριακή κρίση αποτέλεσε ακριβώ το σύμβολο της ίδιας της, της της Ευρώπης να καταπολεμήσει την οικονομική κρίση. Αυτό είναι και το δεύτερο σημείο μου. Δηλαδή θα θέλαμε η Ευρώπη, το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών να προχωρήσουν στο όνομα των πολιτών για αυτά τα ζητήματα των εγγύσεων των καταθέσεων. Αν δεν το καταφέρουμε, δεν το πετύχουμε αυτό μεταξύ μας, τότε η Τραπεζική Ένωση δεν θα γίνει ποτέ αντιληπτή και δεν θα αποτελέσει ποτέ ένα πλεονέκτημα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τρίτο σημείο. Για αυτά που μένουν να κάνουμε για τη ρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα. Αυτοί που ενδιαφέρονται για τα χρηματοοικονομικά διαβάζουν έγγραφα τις τελευταίες εβδομάδες για τους κινδύνους που και πάλι αντιμετωπίζει ο κόσμος και ιδιαίτερα η Ευρώπη. Τι διαβάζουμε. Διαβάζουμε ότι υπάρχει μια φούσκα η οποία ποτέ δεν ε, αντιμετωπίστηκε από τους μηχανισμούς κρίσης μετά το 2008 μια φούσκα χρέους το, δημόσιο, το ιδιωτικό χρέος έγινε δημόσιο η απομόχλευση αυτή η φούσκα λοιπόν δεν έχει τελειώσει οι μηχανισμοί λοιπόν που υλοποιήσαμε στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης μας παρέχουν όμως και χαιρόμαστε γι' αυτό τα μέσα για να προλάβουμε τους ε, κινδύνους που σχετίζονται με αυτά. Όμως, όμως τα έγγραφα αυτά μας λένε ή τα κείμενα αυτά μας λένε ότι υπάρχει ακόμα κίνδυνος για την Ευρώπη. Οι μηχανισμοί διαχείρισης ενεργετικής και παθητικής, δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί παράλληλα ή στο περιθώριο των τραπεζικών μηχανισμών ή κάποιοι Κάποιε τράπεζε απέλεξαν να μην τα περιλάβουν αυτά στου ολογισμού. Αυτό που ονομάζουμε σκιώδη τραπεζική, shadow banking. Έχουμε λοιπόν ε, ε, ασφαλή ζωή, τσάξιο ταμεία και άλλα ταμεία τα οποία αντιμετωπίζουν έτσι κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες και βρίσκονται υπό την επίβλεψη των αγορών. Και εδώ καταλήγω. εμεί έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ για την ρύθμιση των τραπεζών και την υποπτία. Θα πρέπει να κάνουμε το τελευταίο βήμα ώστε να διασφαλίσουμε η τραπεζική αυτή να είναι υπέρ των πολιτών με την, κατα... με την εγγύηση των καταθέσεων. Όμως εμείς ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με μια νέα οικονομική κρίση. Αν αυτή η οικονομική κρίση δεν αφορά μόνο τις τράπεζες αλλά το σύνολο της ε, χρηματοπιστικής αγοράς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Καρίν Μπερζέρ. Να δώσω τώρα το λόγο στην τελευταία ομιλήτρια, τη συνάδελφό μου στην Ολλανδική Γερουσία, την κυρία Ρέτε Πράστα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ συνάδελφε Μάρτιν Φανερόιεν. Σήμερα το απόγευμα μιλώ εκ μέρους της Ολλανδικής Γερουσίας, ε, της οποίας είμαι μέλος ε, ως ε, και εδώ έχουμε μία πρόταση για ένα ευρωπαϊκό ε, σχέδιο εγγύησης καταθέσεων. Ε, λόγω της επιθυμίας να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο σύστημα έχουμε μια διάσταση απόψεων αυτή τη στιγμή στην Ολλανδική Γερουσία και στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Πέραν αυτού όμως θα ήθελα να συζητήσω μια συγκεκριμένη πτυχή αυτού του συγκεκριμένου σχεδίου το ε, Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων. Ένα ε, σχέδιο ασφάλισης καταθέσεων έχει δύο στόχους. Να προστατεύσει τους καταθέτες σε περίπτωση που πτωχεύσει η τράπεζά τους και να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα ε, οικονομικής αστάθειας, ε, κυρίως λόγω bankrun. Προκειμένου όμως να λειτουργήσουν αυτά, θα πρέπει το πρόγραμμα να πληρεί συγκεκριμένε απαιτήσει, διότι η δάλος μπορεί να, μην, να αποβεί βάρος όλων χρειάζονται αλλαγές ε, στην πρόταση, διότι μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Η πρώτη μου παρατήρηση αφορά τις ε, επενδύσεις ε, του Ταμείου. Στην περίπτωση που το Ταμείο θα πρέπει να κάνει πληρωμές ε, στους καταθέτες, ε, τους ε, πελάτες της τράπεζας Υποπτώχευσης, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα ε, χωρίς κόστος. Επομένως, το λογικό θα ήταν το Ταμείο να είναι σε συγκεκριμένο λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, το άρθρο 75.3 της σχετικής πρότασης λέει ότι το Ταμείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για επενδύσεις και ότι θα πρέπει να επενδύεται το κονδύλιο σε υψηλά ρευστά στοιχεία ενεργητικού υψηλής πιστοτικής αξίας. Και φυσικά ε, μιλώ εδώ και εκ μέρου των ε, ε, συναδέλφων γερουσιαστών και σας ζητώ να αποκλείσετε τη δυνατότητα τα κονδύλια του Ταμείου να επενδύονται είτε εμέσως είτε αμέσως σε δείκτες του χρηματιστηρίου, μέσω μάλλον του χρηματιστηρίου, σε τράπεζες οι οποίες περιλαμβάνονται στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων διότι δεν θα θέλαμε να πέσει η αξία του ταμείου την ίδια στιγμή που θα κληθεί να δράσει και να πληρώσει. Και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του ταμείου να πουλά τραπεζικές μετοχές όταν οι τράπεζες ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτό απλώς ε, θα αμβλύνει και άλλο το πρόβλημα. Τώρα, Τρίτο σχόλιο. Αυτό αφορά την περίπτωση στην οποία το Ταμείο θα έχει επιτύχει το στόχο του. Όπως ε, έχει πρόταση αυτή τη στιγμή, από εκείνη τη στιγμή και πέρα, οι τράπεζες δεν θα πρέπει να κάνουν οποιαδήποτε περαιτέρω συνεισφορά. Θυμηθείτε εδώ ότι ε, οποιαδήποτε εισφορά έχει ε, σχέση με κίνδυνο. Αν σταματήσει λοιπόν κάποιος να συνεισφέρει, σταματά να έχει και ε, κάτι το οποίο σχετίζεται με τον κίνδυνό του. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα μπορούν να λαμβάνουν περισσότερου κινδύνους από εκείνο το σημείο και πέρα, διότι δεν θα ε, τιμολογείται αυτό ε, σε ένα υψηλότερο premium που θα έχει στοιχεία κινδύνου. Θα υπάρχει λοιπόν ουσιαστικά ε, ένα στρεβλό αποτέλεσμα, διότι θα ε, επιδοτούμε επικίνδυνες τράπεζες. Αυτό θα επιτρέπει ε, να συνεισφέρουν από τη στιγμή που έχει επιτύχει το στόχο του το Ταμείο επί τη βάση του προφίλ κινδύνου τους εκείνη τη στιγμή, ενώ θα λαμβάνουν μερίσματα βάσει της προηγούμενης συνεισφορά τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε τράπεζες οι οποίες ε, θα ε, είναι πιο ασφαλείς αν πληρώνουν λιγότερο και τράπεζες που θα είναι πιο επικίνδυνες αν πληρώνουν περισσότερα. Αυτέ είναι οι απόψει των εμπειρογνωμόνων μα και των υπολείπων συναδέλφων για τα θέματα αυτά. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία ε, Ριέτ Πράστ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους πέντε ομιλητές ε, ε, για το θέμα αυτό, κυρίως την Ντανιέλ Νιουή και την Έλκε Κένιγκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γουαλτιέρη, ο οποίος θα προεδρεύσει το δεύτερο τμήμα αυτής της συνεδρίασης. Ευχαριστώ. Πρώτος ομιλητής, θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια ε, συνταγή με το πρώτο τμήμα της συνεδρίασης, ο Στέφαν Ράντου Απρέα από τη Ρουμανική Γερουσία. Δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η άποψή μας είναι πως θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή ε, Οικονομική Ένωση, να ολοκληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση μέσω της Τραπεζικής Ένωσης ε, με έναν τρόπο διαφανή που θα περιλαμβάνει τους ε, πάντες και τα 28 κράτη-μέλη χωρίς επιπρόσθετους φραγμούς για τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο ευρώ. Τα απαραίτητα μέσα για την εποπτεία και την διάσωση των τραπεζών υπάρχουν εντός των υφιστάμενων μηχανισμών. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους ε, κανόνες που υπάρχουν μεσοπρόθεσμα πριν ε, φτιάξουμε νέα μέσα. Και οποιαδήποτε νέα μέτρα προβλεφθούν θα πρέπει να αναλυθούν στο πλαίσιο της ευρύτερης ε, εσωτερικής συνοχής, λαμβάνοντα υπόψη βεβαίως και την κυριαρχία των κρατών μελών στα φορολογικά. Παρά το ότι δεν είμαστε μέσα στο ευρώ συμμετείχαμε στην ε, διαμόρφωση ακριβώς της Τραπεζικής Ένωσης και της εποπτείας του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Σας ευχαριστώ. Τώρα ο Χάνς Μίκελμπαχ από την Γερμανική Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ ακόμη μια φορά στα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια όσον αφορά τις ε, τραπεζικές ε, μετοχές, κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με την Τραπεζική Ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί ο τραπεζικός τομέας ε, είναι τώρα καλύτερα διαχωρισμένος από την υπόλοιπη οικονομία χάρη σε ενέργειές μας μέσω της ε, Τραπεζικής Ένωσης, αλλά πολλοί επενδυτές εξακολουθούν να έχουν προβλήματα εμπιστοσύνης και συνειδητοποιούν πως κάποιες τράπεζες δεν είναι τόσο υγιείς ε, και το θέμα είναι πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και βεβαίως βλέπουμε πως κατά την άποψή μου φταίει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ πέρα και οι κεντρικές τράπεζες οι οποίες με την ε, ποσοτική νομισματική χαλάρωση εμπόδισαν ή καθυστέρησαν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και έδωσαν απεριόριστο φτηνό χτήμα στις ε, τράπεζες και δεν χρειάζεται να αναζητήσουν επιπλέον ρευστότητα. Λόγω λοιπόν της περιορισμένης σχετικά κεφαλαιακής τους ε, βάσης, οι ευρωπαϊκές τράπεζες ε, στην διεθνή σύγκριση εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ ασθενείς και αυτό δυστυχώς ε, δεν ωφελεί και την πραγματική ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό θα λυθεί οπωσδήποτε βέβαια στο μέλλον με την Τραπεζική Ένωση, αλλά αυτή τη στιγμή οι δυσκολίες που έχουμε ε, είναι ένα ζήτημα το πώς θα το αντιμετωπίσουμε ειδικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στα χρηματιστήρια. Είναι πολύ βασικό αυτό. Σας ευχαριστώ. Ενρίκο Δίας ε, από την Πορτογαλική Βουλή. Ε, ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς γιατί για τις πολύ καλές εισηγήσεις που ακούσαμε που συμβάλλουν θετικά στη συζήτηση και είναι πολύ χρήσιμες. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που θεωρώ σημαντικά στα πλαίσια αυτών των δύο λεπτών. Καταρχάς αυτή η έλλειψη ισορροπίας που έχουμε στην Τραπεζική Ένωση δηλαδή το γεγονός ότι ο τρίτος πυλώνας δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα αυτό το γεγονό κάνει κάποιε χώρε μέλη να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ω ψηλότερο από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Και κάποιε επιχειρήσει πληρώνουν περισσότερο ε, μέσω των spread για αυτό το κίνδυνο. Αυτό νομίζω στρεβλώνει την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό. Οπότε αυτά που λέμε για την εγγύηση των καταθέσεων είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, η πολύ εύθραυστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται κάποιες τράπεζες. Είχαμε διαδικασίες εξυγένσης ε, τραπεζών όπως οι πορτογαλικές που ήταν στα παρουσία των εφημερίδων. Ακούμε τώρα ότι υπάρχει μια διαδικασία συγκέντρωση και αυτή η διαδικασία νομίζω είναι επικίνδυνη γιατί ακριβώς προσπαθούμε να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα σύνολο τραπεζικών οντοτήτων μεγάλων διαστάσεων που είναι υπερβολικά μεγάλες για να πτωχεύσουν. Αυτή η διαδικασία λοιπόν μα φαίνεται κάπω επικίνδυνη. Αντίθετα, σε άλλε χώρες όπως είπα, ο κατακαιρματισμός ακριβώς του τραπεζικού τομέα κάνει ελέξιμες και διαχειρίσιμες αυτές τις καταστάσεις, στόχες δηλαδή μεγάλων τραπεζών ή ιδρυμάτων. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις ε, τράπεζες οι οποίες στην Ευρώπη είναι υπερβολικά μεγάλες για να πτωχεύσουν. Και ένα τελευταίο. Οι εμπορικέ τραπέζες θα πρέπει να διαχωρίζονται από τις ε, επενδυτικές τράπεζες. Γι' αυτό το θέμα θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Δική Πρόεδρος. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ελίζα Φερέρα, σκιώδης συζητητής και αυτή για αυτό το θέμα εγγύησεων καταθέσεων. Ναι, θα μιλήσω αγγλικά, δεν κύριε Φερέρα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήρθατε εδώ και για την συνεχή δουλειά που κάνετε. Έχουμε δύο γυναίκες οι οποίες ηγούνται αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλες τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, αλλά και για το γεγονός ότι συνεχίσατε τις επαφές με το Κοινοβούλιο. Οι ερωτήσεις μου και οι αμφιβολίες μου έχουν θετικό χαρακτήρα και επικοδομητικό, επειδή νομίζω το Κοινοβούλιο ήταν πραγματικά επικοδομητικό στην εικασία αυτή. Για τις λεπτομέρειες αυτής της μετάβασης από μια κοινή προσέγγιση για τα τραπεζικά θέματα σε μια νέα φάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Τραπεζική Ένωση γιατί εσείς έχετε ουσιώδη ρόλο στην δημιουργία αυτού του νέου πλαισίου αυτής της νέας υποδομής η κυρία Κένινγκ προηγουμένω είπε ότι ο στόχος σας δεν είναι το να έχουμε εξυγένση τραπεζών, αλλά να αποφύγουμε την εξυγένση. Ταυτόχρονα όμως, ήδη προκαταλαμβάνουμε κάτι το οποίο είναι η BRD. Η πρώτη φορά είναι που γίνεται στην Ευρώπη αυτό. Και ακόμα δεν το έχουμε δοκιμάσει, δεν είναι δοκιμασμένο, σε μεγάλο ποσοστό. Αυτό ήδη εφαρμόζεται, αλλά εφαρμόζεται πριν ολοκληρώσουμε το σύνολο της δομής που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Πριν δηλαδή υποφερθούμε από τις θετικές επιπτώσεις στην αγορά. Λείπουν κάποια στοιχεία, λείπουν ας πούμε η κοινή γραμμή, το DGS, που και αυτό λείπει Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα κίνδυνο. Η εφαρμογή της BRRD να βρεθεί στα πλαίσια ενός συστημικού κινδύνου και όπως είπε και ο Γερμανός συνάδελφος τι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις και όπως είπε και ο Πορτογάλος συνάδελφος ο συμπατριώτης μου μαζί με τις αρχές του ανταγωνισμού και την Κομισιόν προσπαθείτε να βρείτε έτσι μια εικόνα, ένα όραμα για κάθε χρηματοπιστική αιρώα, ώστε να υπάρξει σύγκληση σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Στενέκ Βέστα από τη Ρουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Δεν θα μιλήσω τεχνικά. Να πω μόνο ότι υπάρχουν τράπεζες στην Ένωση που είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Έχουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία. Άλλες τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα και βρίσκονται σε φάση και εκαθάρισης. Είτε επειδή οι πελάτες δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους ή επειδή ακολούθησαν ασφαλμένες πολιτικές. 700 εκατομμύρια κορώνες, 28 εκατομμύρια δηλαδή ευρώ. Αυτό θα πρέπει να δώσει, έπρεπε να δώσει η Τσεχική αυτο θα πρεπει να δωσει επρεπε να δωσει η τσεχη δημοκρατια στις τράπεζες και τώρα τα χρήματα μας λείπουν. Τώρα οι τράπεζες είναι σχετικά υγιείς, τουλάχιστον έτσι λένε αυτές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλες αυτές οι τράπεζες είναι θηγατρικές μεγάλων πολυεθνικών τραπεζών και εδώ ακριβώς υπάρχει ο κίνδυνος ότι ε, σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση οι τράπεζες όταν θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν τα χρήματα από τις υγιείς θηγατρικές προς τις μη υγιείς θηγατρικές σε άλλες χώρες. Οπότε θα ήθελα εγώ να μάθω η Τραπεζική Ένωση έχει μια πρόβλεψη και διαθέτει επαρκή εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, να αποφύγουμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι νομίμο αλλά δεν είναι ηθικό γιατί στην ουσία αποτελεί επιδότηση κάποιων τραπεζών εις βάρος κάποιων άλλων. Και χάρηκα που άκουσα για το BEPS, χάρηκα που θεσπίστηκε αυτό ως πλαίσιο αλλά θα πρέπει να έχουμε και μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν σε μια πανευρωπαϊκή οικονομική σταθερότητα. Είτε πρόκειται για την εγγύηση των καταθέσεων, είτε για τον BEPS, είτε για την εποπτεία. Όλα είναι ευπρόσδεκτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φρανσουά Μάρ από την Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ. πρέπει να προχωρήσουμε σημαντικά για την ε, τραπεζική ε, ρύθμιση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτά τα οποία διευκρινίστηκαν προηγουμένως στην εισαγωγή και να ευχαριστήσω και τους ομιλητές για τις διευκρινήσεις που μας έκαναν. Ωστόσο, εξακολουθούμε να έχουμε ανησυχίες. Η πρώτη αναφέρθηκε μόλις προηγουμένως, το πόσο ευμετάβλητο είναι το χρηματιστήριο όσον αφορά τους ε, τραπεζικούς τίτλους και το είδαμε και τις τελευταίες ημέρες με πολύ σημαντική πτώση για κάποιες τράπεζες στην Ευρώπη. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο επισημάνθηκε είναι το θέμα του κινδύνου και να ευχαριστήσω την Red Πράστ που ε, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό ε, πολύ εύστοχα. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις όσον αφορά τη ρύθμιση και την έκταση που θα πρέπει να λάβει. Επίσης, ε, κυρίως όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες ε, που διεξάγουν οι τράπεζες εκτός του ισοζυγία τους, δηλαδή όλο αυτό το shadow banking, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα για το οποίο σχολίασαν και οι παρατηρητές και οι θύνοντες ότι πρέπει να εποπτεύουμε για τον σχετικό κίνδυνο όλων αυτών των διαδικασιών. Και το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η συνοχή ε, των μέτρων ρύθμισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά τις πολιτικές ε, ε, ρύθμισης και εποπτείας που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Και σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, όπως και αρκετοί άλλοι, έμαθα ε, τη δήλωση του Τζον Βίκερς που γνωρίζουμε ότι είναι ένας από τους ε, ε, γυρεότερους και μπόρεσε να συνεισφέρει πάρα πολύ στα θέματα της Τραπεζικής Ένωσης. Υπάρχει ένα άρθρο στον τύπο που λέει σήμα κινδύνου για την τραπεζική ρύθμιση στην Ευρώπη και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα να ξέρω αν γνωρίζετε ε, κάτι σχετικά ε, με το σημείο αυτό. Τι άποψη έχετε εσείς επ' αυτού για τις ε, παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι είναι αρκετά ικανοί να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα τραπεζικά αυτά ζητήματα. Τι άποψη έχουμε λοιπόν εμείς σήμερα για αυτό το σήμα κινδύνου που στέλνουν προσωπικές κότητες όπως ο κύριος Βίκερς. Ευχαριστώ ο Φραντσέσκο Καριέλο από την ε, Βουλή της Ιταλίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το Ιταλικό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα το οποίο δεσμεύει την κυβέρνηση για την αναστολή του Μπέιλιν. Το Κοινοβούλιο πρότεινε ένα ψήφισμα το οποίο υπέβαλε η αντιπολίτευση. Μία μικρή μειοψηφία στην ε, Ιταλική Βουλή πιστεύει ότι θα πρέπει να ανασταλεί επαόριστον η όλη διαδικασία διάθεση των τραπεζών εδώ. Εγώ εκπροσωπώ αυτή τη μειοψηφία και πρέπει να σας πω ότι το όραμά μας ε, πηγαίνει σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από ε, το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι δεν αποτελεί λύση ε, η συγκέντρωση των τραπεζικών δυνάμεων για τα τραπεζικά προβλήματα, γιατί υποδα... σκάπτουν ε, την δημοκρατία των χωρών και την ανεξαρτησία του τραπεζικού συστήματος. Διότι ε, το να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε σε μεγάλους πόλους το τραπεζικό σύστημα σημαίνει ότι θα καθορίζουμε και την πολιτική των κυβερνήσεων. Όπως έλεγα λοιπόν, η άποψή μας είναι η εκ διαμέτρου αντίθετη. Εμείς είμαστε υπέρ του διαχωρισμού των εξουσιών και των τύπων ε, τραπεζών, από τις εμπορικές τράπεζες ε, και ε, τις υπόλοιπε κατηγορίες και πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε μία σαφή και προφανή γραμμή που πηγαίνει προς την συγκέντρωση των χρηματοπιστωτικών εξουσιών. Και αναρωτιέμαι και θα ήθελα να ρωτήσω και τους παρισταμένους. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι όντως με τους πολίπες, έχει, έχει μία απόφαση κατά του Ευρωπαϊκού Μονοπωλίου που είχε δημιουργήσει ένα καρτέλ ε, με τα Euribor και τον καθορισμό των επιτοκίων του Euribor. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση διάφοροι καταναλωτές και καταθέτες θα μπορούσαν να καταγγείλουν και να επικαλεστούν τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση για να αποζημιωθούν για ένα ε, για μια υψηλού επίπεδου πάτη από αυτά τα καρτέλ των τραπεζών όπως η Barclays, η Deutsche Bank, και η Royal Bank of Scotland ε, και θα ήθελα να ξέρω προς ποια κατεύθυνση οδεύουμε. Είμαστε με το μέρος των πολιτών ή όχι. Indeed, the text of the resolution. Σας ευχαριστώ. Πράγματι ήταν κάπως διαφορετικό το κείμενο του ψηφίσματος, αλλά όλοι έχουν τις απόψεις τους. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε τον λόγο τις ε, κυρίες Νίγη και Κένικ για κάποια σχόλια. Ακούσατε πολλές ερωτήσεις, ε, κάποιες συγκεκριμένες, κάποιες ε, δύσκολες. Παρακαλώ. Λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, θα πρέπει να είμαι πολύ γρήγορη. Και βεβαίως θα αφήσω τις υπόλοιπε που δεν με αφορούν για την κυρία Κένιγκ. Δεν ναι, βλέπω τώρα πως ε, μας ε, ζητήσατε για την ε, οδηγία να επιδείξουμε κάποια ευελιξία γιατί υπάρχουν και κάποιες ασάφειες όσον αφορά το μέγιστο πόσο διανομής αλλά όταν καλυφθεί αυτό μετά δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο ευελιξίας το μέγιστο ποσό διανομής είναι σαφές, ξεκαθαρό και καλύπτει και τη διανομή μερίσματος που δεν χρειάζεται τόσο πολύ κατά την άποψή μας γιατί είναι το, το, το μέγιστο μόνο και ήδη χρησιμοποιούμε ε, σκληρούς ε, κανόνες ε, γι' αυτό αλλά και κουπόνια επίσης τα οποία αποπληρώνονται με άλλα μέσα tier 1 επίσης οφείλονται στο ότι οι αγορές χωρίς το κουπόνι δεν αντιλαμβάνονται δεν ξέρουν ότι θα υπάρξει κάποια εξόφληση την στιγμή που πρέπει οπότε υπάρχει κάποιος κίνδυνος και βέβαια αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο θα λάβουν κάποια μπόνους και κάποια αποσημείωση που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από μερίσματα και κουπόνια κτλ. Οπότε θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσει ε, όσον αφορά τον κανονισμό. Το άλλο θέμα αφορούσε την έκθεση σε κρατικό χρέος. Συμφωνώ πως η τελευταία αυτή η οικονομική κρίση έδειξε πως η έκθεση κρατικό χρέος δεν είναι χωρίς κείμενο, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν κεφαλαιακές απαιτήσει. Προφανώς αυτό πρέπει να γίνει προσεκτικά και γνωρίζουμε πως γίνεται κάποια δουλειά σε διεθνές επίπεδο, οπότε καλύτερο είναι να μην προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια ενιαία ευρωπαϊκή ε, λύση, σε ένα ζήτημα το οποίο είναι διεθνές θα έχουμε παραδείγματο χάρη την πρόταση της Επιτροπής της ε, Βασιλείας πρώτα και μετά θα αποφασίσει η Κομισιόν πώς θα την εφαρμόσει. Όσον αφορά τώρα τον πυλώνα που λείπει από την Τραπεζική Ένωση, συμφωνώ απολύτως με αυτούς που το είπαν και αυτό ακριβώς λείπει από την Τραπεζική Ένωση. Θα προσθέσω πως χρειάζεται και μια δημοσιονομική λύση ανάγκης για το ενίο ταμείο διάσωσης. Θα σταματήσω εδώ για αυτό το θέμα. Και προφανώς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, ε πολιτική της ε, Οικονομικής Ένωσης για να μπορούν οι αποδομευτές να εμπιστευτούν τα λεφτά τους στις τράπεζες. Επίσης κάτι υπόθηκε για την Πορτογαλία για την πιθανή συγκέντρωση σε δύο μεγάλες ε, τράπεζες. Ε, κοιτάξτε, εξαρτάται από την κάθε χώρα. Σε κάποιες χώρες είναι πολύ συγκεντρωμένα τα τραπεζικά συστήματα και δεν υπάρχει άλλο περιθώριο συγχωνεύσεων, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όπου ε, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία και ίσως υπάρχει περαιτέρω περιθώριο κάποιων συνενώσεων. Σε κάποιες χώρες αυτό θα συμβεί τώρα για το εάν συνεργαζόμαστε στενά με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ναι, όντως. Και πράγματι εδώ πέρα πράγματι έχει αλλάξει η κατάσταση γιατί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνεννοούνται μεταξύ τους ε, εδώ πέρα δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση με τη Γενική Διεθνή συνταγωνισμού, για την ερώτηση του Τσέχου βουλευτή αν δεν κάνω λάθος για το εάν αποτρέπουμε επιδοτήσεις διαφορετικών κομματιών ενός ομίλου. Κοιτάξτε, στόχος είναι να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός. Θέλουμε εντός της Τραπεζικής Ένωσης να θεωρούμαστε μια ενιαία εποπτική αρχή, να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων και είμαστε υπερήφανοι για το ότι θεωρούμαστε ε, έτσι από τα stress test της ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής που στόχο έχουν να καλύπτουν το 70% των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών σε κάθε χώρα. Το πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης, κάτι το οποίο οπωσδήποτε δίνει έμφαση στις μεγαλύτερες χώρες ε, που είναι λογικό νομίζω. Όσον αφορά την ε, ρύθμιση των τραπεζών και αυτά τα οποία ε, υπόθηκαν για το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχω άποψη δεν ξέρω, ίσως είναι ευκαιρία να δώσω τον λόγο στην ε, κυρία Κένιγκ εδώ πέρα. Γιατί όσον αφορά την αναβολή της εφαρμογής ε, του κανονισμού του bail-in, δεν ξέρω αν καλή ιδέα, γιατί σταδιακά οι αγορές συνηθίζουν στην ιδέα, έχουν αντιληφθεί πως ε, από πρώτης πρώτου φέτος είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και η μεταβατική περίοδος πάντα είναι πιο ευαίσθητη και λεπτή, αλλά νομίζω πως πολλά έχουν ήδη γίνει για να γίνει σωστά αυτή η μετάβαση. Η κυρία Κένιγκ, σας ευχαριστώ. Νόμιζα πως η Ντανιέλ μου έδωσε τον λόγο να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σεβίκτης, γιατί και εγώ δεν θα ήθελα να απαντήσω. Να αναφερθώ στο τελευταίο σημείο Κοιτάξτε, νομίζω πως πάει μακριά να συνδέσουμε την θέση ενισχύ της οδηγίας BRD με την ε, τωρινή κρίση. Εγώ θα πω αυτό το οποίο είπα, διάβασα χτες τους Financial Times ότι ο κανονισμός ε, de minimis για τα επιέλατων είναι πίσω σε ένας ύποπτος αλλά τώρα υπάρχει αυτή η οδηγία και πρέπει να την εφαρμόσουμε. Είναι λοιπόν ένα μηχανισμό ο οποίο ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ενιαίο μηχανισμό διάσωση επίση. Πρέπει να είμαστε συνεπεί, προβλέψιμοι στο πώ ε, δρούμε και να υπάρχει διαφάνεια. Οπότε το να λέμε μόνο ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό βεβαίω. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη πως ε, σε κάποια κρατημέλη υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα και πρέπει να ε, δρούμε αναλογικά και με την κατάσταση. Αλλά να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε η Ντανιέλ. Υπάρχει λίγο αυτό το σκεπτικό το ότι μήπως ενθαρρύνουμε έτσι την συγκέντρωση στην αγορά. Δεν είμαι σίγουρη ότι συμφωνώ τόσο. Βεβαίως ε, υπάρχει σε μια αγορά κάποια συγκέντρωση, αλλά βλέπουμε επίσης πως οι τράπεζες χωρίς ε, κάποιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο κάποια στιγμή θα πρέπει να ε, οδηγηθούν σε αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή ότι αλλάζει το παιχνίδι, να έχουν κάποια ευρωστία που θα τους επιτρέψει να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Επίσης είπατε πως πρέπει η Τραπεζική Ένωση να είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη-μέλη, οπωσδήποτε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Σαφώς είναι ένα βήμα το οποίο πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη και εγώ είπα στην αρχή πως εγώ θα πω πως ε, είναι νίκη για την Τραπεζική Ένωση αν σκεφτεί και το Ηνωμένο Βασίλειο να ενταχθεί. Ε, για την ώρα πάντως είναι ανοιχτό για όλα τα κράτη-μέλη, αυτό είναι σαφές. Υπήρχαν σχόλια για την σκιώδη τραπεζική, εμείς πάντα λέγαμε πως θα πρέπει η ρύθμιση να είναι διάφανη και να μην υπάρχει δυνατότητα κάποιος να επιλέγει εντός του συστήματος. Αλλά τέλος δεν θα το, επιλέγει, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς αυτό τώρα. Έγιναν κάποια πολύ συγκεκριμένα σχόλια. για το TGF και τις επενδύσεις ε, εκεί υποθέτω πως ε, θα έχουμε παρόμοιους κανόνες με το ε, ενίο ταμείο διάσωσης και θα συμφωνήσω πως ε, ίσως δεν είναι τόσο καλή ιδέα να επενδύει κανείς σε αυτούς που μετά θα πρέπει να διασώσει. Και μιλήσατε για κάποια επίπεδα στόχο στο μέλλον. Και ελπίζω ο νομοθέτης να το λάβει αυτό υπόψη. Και πάντα έλεγα πως σαφώς η Τραπεζική Ένωση έχει τρεις πυλώνες, τρία σκέλια, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να αποκτήσουμε κάποτε ένα εναρμονισμένο σύστημα εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και να εναρμονιστεί ακριβώς αυτή η σχέση μεταξύ των εθνικών συστημάτων και του ταμείου, των εθνικών συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και του Ταμείου Διάσωσης και μετά έρχομαι σε αυτό το οποίο είπε η Ντανιέλ. Να μην ζητήσουμε δηλαδή ταυτόχρονα και εναρμόνιση του ε, δικαίου, του πτωχευτικού, αλλά να μην παραμελούμε και τα εύκολα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Παραδείγματο χάρη μια ιεράρχηση των πιστωτών ή τους ε, τομείς ε, αναποτελεσματικής λειτουργίας κάποιων εθνικών συστημάτων χρεοκοπίας οπότε μετά το Ταμείο Διάσωσης να είναι το μόνο το οποίο θα έχει τα μέσα για να αγγίθει τις καταθέσεις κτλ. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν που πρέπει να γίνουν και δεν θα αλλάξουν δραματικά την κατάσταση αλλά πρέπει να γίνουν σιγά σιγά και επίσης όταν μιλήσατε για κάποιο, κάποια δημοσιονομική λύση ανάγκης ναι, ας υπογραφούν όλα αυτά και μετά έχουμε και άλλη δουλειά που πρέπει να γίνει. Thank you very much. I think... Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργεία νομίζω. Πολύ σημαντικά ζητήματα συζητήσαμε. Να ευχαριστήσω και πάλι την Δανιέλ και την Έλκη. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε βέβαια με τα πάντα 100% πάντα θα υπάρχει διαφορά σε αφορά το περιθώριο επιλεξίας του MDA αλλά πάντως χαιρετίζω το γεγονό ότι αναγνωρίζετε ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις όσον αφορά τα προβλήματα της αγοράς 81. Θα σκεφτούμε λοιπόν τι λύσεις μπορούμε να βρούμε στα διάφορα προβλήματα και χαιρετίζουμε και αυτά που υπόθηκαν για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Βέβαια υπάρχει μια νομοθετική διαδικασία που δεν θα αναφέρουμε λεπτομερώς, αλλά υπάρχει θετική στάση. Και συμφωνώ με την Έλκε και Νίκ ότι η αναβολή ενός πράγματος που έχει τεθεί σε ισχύ δεν έχει νόημα και συμφωνώ με αυτά που είπατε για την αναλογικότητα που αφορά τη σταθερότητα την οικονομική. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και είναι σημαντικό αυτό που είπατε σχετικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τις δύο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φαντρόν στον συμπρόεδρο, ο οποίος λέει ότι θα ήθελα ε, εκ μέρους του συναδέλφου Ετσίνκα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές των δύο συνεδριών που μίλησαν για την Τραπεζική Ένωση. Να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες για αυτές τις δύο συνεδρίες και από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό και λύνουμε αυτόν τον τρόπο την τελευταία συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ.